Sí, buenos días a todos. Yo pido que vayan tomando... Καλημέρα Σα παρακαλώ καθίστε σιγά σιγά γιατί δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε περισσότερο την έναρξη του εργαστηρίου workshop γιατί έχουμε και άλλα σημεία κατά τη διάρκεια της που πρέπει να εξετάσουμε. Λυπούμε γι' αυτό. Καλωσορίζω όλου του προσκεκλημένους που έχουμε για το εργαστήριο workshop που όπως ε, γνωρίζετε θα εξετάσει ένα πολύ σημαντικό θέμα τις αλλαγές καθεστώτος στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Μια και δεν είναι πολλοί οι ευρωβουλευτές παρόντες, είναι το αποτέλεσμα μάλλον του χθεσινού ποτού του κοκτέιλ. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει το πράγμα, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Και θα διαρθρώσουμε με τον εξή τρόπο τις εργασίες μας. Κάθε ένας από τους μας θα έχει το μέγιστο 15 λεπτό για την παρέμβασή του. Μετά στο τέλος θα έχουμε 40 λεπτά διαθέσιμα για να έχουμε μια ευρύτερη ανταλλαγή απόψεων μέσας και τους ε, βουλευτές. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε με τον δόκτορα κύριο Κρίστιαν Μέλμαν από το Ίδρυμα Ιδροβιολογίας και Αλίας ε, του Πανεπιστημίου του Αμβούργου. Θα μας μιλήσει για το καθεστώς των οικοσυστημάτων και τις αλλαγές ε, όσον αφορά την υπεραλίευση. Ο κύριος ε, Δόκτωρ Μέλμαν έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Για 15 λεπτά κατά το μέγιστο. Ευχαριστώ. Should I start? okay. Εντάξει. Καλή σα μέρα λοιπόν. Τα οικοσυστήματα και οι επιπτώσεις ε, της υπεραλίευση. Μία αναθεώρηση με μεγάλων μελετών όσον αφορά αυτές τις αλλαγές στο Βορείο Ατλαντικό Και προτού ξεκινήσω με αυτή την επισκόπηση, θα ήθελα να δώσω τον ορισμό των αλλαγών και μεταβολών οικοσυστημάτων ε, γιατί πολύ συχνά χρησιμοποιείται και δεν χρησιμοποιείται πάντα σωστά και η μελέτη που έχουμε εδώ όσον αφορά τις αλλαγές καθεστώτος χαρακτηρίζονται σε σχέση με την συχνότητά τους. Δεν είναι υπερβολικά συχνές αυτές, αλλά είναι απότομες, αυτό είναι το πιο σημαντικό, απότομες περίοδοι αλλαγών όσον αφορά τις μεταβολές αυτές σε σχέση με τα καθεστώτα των οικοσυστήματων. Σημαντικό για την δική μου επισκόπηση είναι εξετάζω αυτές τις αλλαγές και τις δομές σε σχέση με τη μελέτη αυτή και τα όσα εξέτασα στο σύνολο των οικοσυστήματων από το πλανκτόν μέχρι και τις, τα, τα ε, ψάρια κυνηγού και τις αλλαγές σε μεγάλη κλίμακα, δηλαδή την μεγάλη κλίμακα οικοσυστημάτων, για παράδειγμα το Βορειοατλαντικό, την ε, Βαλτική, Μαύρη Θάλασσα κλπ. που περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Συνοψίζω λοιπόν, έχουμε τα, τις κυριότερες αλλαγές ε, στα οικοσυστήματα και τα κυριότερα αίτια και σε, ένα δεύτερο, ε, σε μια δεύτερη φάση αναζητούμε το, ε, να βρούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις της υπεραλίευσης, πώς αυτή μπορεί να προκαλέσει αυτές τις αλλαγές ε, στο ε, θαλάσσιο οικοσύστημα, στην τροφική αλυσίδα. Και μ, ξεκινώ με αυτόν τον τρόπο, διότι θεωρητικά αν αυτά τα καθεστώτα είναι σταθερά, σε σχέση με την διαχείρισή τους και τις επιπτώσεις, που υπάρχουν παρουσιάζω κάποια συμπεράσματα για τις, ε, τα αίτια των ε, μεταβολών αυτών στα οικοσυστήματα λόγω υπεραλήψης και στο τέλος ε, εξετάζω τις επιπτώσεις για τη διαχείριση αλλά όχι υπερβολικά, στη συνέχεια θα ακολουθήσουν περισσότερες λεπτομέρειες. why are of... Και οι αλλαγές αυτές αποτελούν αντικείμενο ανησυχίας για τη διαχείριση. Αν δείτε ότι ε, στη φάση τη θεωρητική της εξέτασης των οικοσυστημάτων αντιδρούν σε πιέσεις, σε εξωτερικές πιέσεις όπως αλία για παράδειγμα, την αλίευση και βλέπουμε γραμμικά τις αντιδράσεις όσον αφορά την πίεση που υφίστανται τα οικοσυστήματα, όσον αφορά την υγεία τους ε, με ένα γραμμικό τρόπο. Και μια άλλη δυνατότητα είναι στην κόκκινη γραμμή για παράδειγμα που έχουμε με την αύξηση των πιέσεων αλλάζουν υπερβολικά μέρση. Και όταν φτάνουμε στο κατόφλι, το κρίσιμο κατόφλι, υπάρχουν απότομες αλλαγές, απότομες αλλαγές ε, κατάστασης. Έχουμε λοιπόν αυτό το κατόφλι που αντιδρά ταχύτατα και απότομα ένα οικοσύστημα. Μετά πρέπει να αναζητήσουμε ένα τρίτο είδος αντίδρασης ε, σε σχέση με την αυξανόμενη πίεση, με την κόκκινη γραμμή, βλέπουμε την αλλαγή που υφίστανται τα οικοσυστήματα και ξαφνικά απότομα, όταν φτάνουμε στο κατόφλι μετά αλλαγών, μπορείτε να δείτε ότι αμέσως υπάρχει η αρνητική αυτή εξέλιξη, παράλληλα με την κόκκινη γραμμή, όμως σε αντιδιαστολή με αυτήν αν αφαιρεθεί η πίεση και υπάρχει η δυνατότητα ανάκαμψης ή επαναφοράς, τότε έχουμε δύο εναλλακτικές προοπτικές σε αυτή τη φάση. Θα μπορούσε είτε να μειωθεί η πίεση, για παράδειγμα, σε σχέση με τη, τον, την αλλιευτική προσπάθεια, ή να περάσουμε σε ένα νέο καθεστώς. Περισσότερες λεπτομέρειες ιστερότερα για αυτά. Αυτές είναι οι, αυτά, αυτό το σκηνικό για τη θεωρία για τις αλλαγές οικοσυστημάτων Πέντε οικοσύστηματα εξετάζω. Με το βόρειο ειρηνικό ξεκινώ στα αριστερά, που θα έλεγα είναι το πρώτο οικοσύστημα που έχει τόσο σε βάθος μελετηθεί σε αυτή τη βάση. Δεύτερον, δυτικός Ατλαντικός και το, τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα, βόρεια θάλασσα, βαλτική θάλασσα, λεπτομέρειες πάλι για αυτά υστερότερα. Επέλεξα αυτές τις μελέτες ε, βασιζόμενος σε κάποια συγκεκριμένα κριτήρια βέβαια που αναφέρονται από πλευρά στους ορισμούς των ε, αλλαγών ε, που προανέφερα και από το τροπικό επίπεδο, τροφικό επίπεδο, πλανκτών, υποπλακτών διότι οι αλλαγές στα οικοσυστήματα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όλες τις αλλαγές στις διαθρώσεις των οικοσυστημάτων συλλήβδη. Και με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία για να αναλύσουμε τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων και χρησιμοποιούμε πολυσχηδή στατιστικά στοιχεία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μελέτες που χρησιμοποιούν μεθοδολογικά ε, προσεγγίσεις που μπορούν να ε, ανακεφαλαιώνουν αυτές τις αλλαγές και ε, περιληπτικά να μπορούμε να τις εξετάσουμε. Και οι απότομες ξαφνικές αλλαγές που και αυτές είναι ένα σημαντικό κριτήριο με ε, μελέτες που έχουν επιλεγεί σχετικά. Αυτά ισχύουν για τα 20, το οικοσύστημα του ε, ειρηνικού. Έχουμε λοιπόν εδώ και το θέμα του Ατλαντικού, Βόρειο Ατλαντικού και Βόρεια Θάλασσα και Βαλτικής Θάλασσα και για την ε, Μαύρη θάλασσα έχουμε αλλαγές που είναι μία από τις καλύτερες μελέτες οικοσυστημάτων και περισσότερες πάλι λεπτομέρειες για αυτό το θέμα Ιστερότερα. Μπορείτε να δείτε εδώ ένα παράδειγμα μια τέτοια μελέτη αλλαγή ε, καθεστώτο. Στο αριστερό πλευρό μπορείτε να δείτε δύο δείκτε ε, που ε, μέσα στη χρονική διάρκεια επισημαίνουν, δείχνουν αυτές τις αλλαγές. Αυτοί οι δείκτες δείχνουν αλλαγές στα οικοσυστήματα. Το πρώτο, ο πρώτος, ο μαύρος, είναι ο δείκτης που δείχνει τις αλλαγές όσον αφορά τις περισσότερες συνιστώσεις ενός οικοστή Ο δεύτερος δείκτης δείχνει αναλογικά ποιες είναι οι αλλαγές ε, του συγκεκριμένου οικοσυστήματος. Βλέποντας αυτά με την κόκκινη διακεκομένη γραμμή, αυτό, αυτή δείχνει πότε αλλάζουν αυτοί οι δείκτες ε, με ταχύτερους ρυθμού. Η πρώτη αλλαγή κατά την, τα μέσα της ε, δεκαετίας του 70 και μετά στη δεκαετία του 80 είναι η χαρακτηριστική περίοδος ε, αυτών των μεγάλων αλλαγών στους ωκεανούς. Ε, και δεξιά βλέπετε αυτούς τους δείκτες ε, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ο ένας με τον άλλο για να συγκρίνουμε τις αλλαγές. Βλέπετε μέσα από το τη χρονική διάρκεια της αλλαγές που επέρχονται στη χρονική κλίμακα στη δεκαετία 60, δεκαετία 70, απότομη αλλαγή κατά τη δεκαετία του 70, νέο καθεστώς που αναδύεται, μετά μια άλλη μεταβολή κατά τα τέλη της δεκαετίας του 80, όπου βλέπουμε ότι με, του, με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια συγκρίσιμη αλλαγή για να παρατηρήσουμε τις χαρακτηριστικές αυτές μεταβολές και στην έκθεση θα βρείτε ότι αυτό ισχύει για όλα τα οικοσυστήματα γενικά. Αν όλα αυτά τα στοιχεία για τα οικοσυστήματα και το καθεστώς τους τα αναφέρουμε σε, αυτό το, σε αυτούς τους δείκτες για τις αλλαγές των οικοσυστημάτων συνολικά, πράγμα που έκανα σε αυτή τη διαφάνεια που βλέπετε εδώ, στη φάση αυτή που συγκρίνει τα οικοσυστήματα μέσα σε μια χρονική διάρκεια βόρειο ειρηνικό, την ε, ε, περιοχή γύρω από τη Δανία, τη Βαλτική θάλασσα. Βλέπετε ότι όλοι αυτοί οι δείκτες έχουν μια συγχρονία στην ε, ανάπτυξη, στην εξέλιξή τους βλέπετε τις αλλαγές από τα μέσα της δεκαετίας του 80 έως τα, στις αρχές της δεκαετίας του 90 από μία έως και περισσότερες φάσεις που βρίσκονται υπό εξέλιξη και αναπτύσσονται. Και σε σχέση με την μαύρη γραμμή βλέπουμε έναν μέσον όρο, έχουμε τα μέγιστα επίσης, τις μέγιστες διακυμάνσεις, έχουμε τους δείκτες για αυτές τις αλλαγές, οι περισσότεροι δείκτες προέρχονται από μια ένα μεγάλο εύρος περιοχών από τις πιο μακρινές περιοχές ε, του Ειρηνικού μέχρι και την ε, Βαλτική θάλασσα από πολύ διαφορετικά οικοσυστήματα συνολικά. Αν επισκοπήσει κανείς ε, τη βιβλιογραφία, πολύ συχνά οι αλλαγές αυτές που από τις κλιματικές αλλαγές. Και έχω εδώ και τους δείκτες αυτούς για τον Βόρειο Ατλαντικό και τις διακυμάνσεις σε αυτόν τον ωκεανό που είναι μια αντανάκλαση των περισσότερων ε, κλιματικών ε, αλλαγών και ε, διαφορετικών συνθήκων που ισχύουν εκεί σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι ένας μια καλή επισκόπηση. Βλέποντας αυτόν τον πίνακα και τις μελέτες που είχαμε αντλήσει αυτά τα στοιχεία, βλέπετε ότι έχουμε κατά τα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές της δεκαετίας του 90 τις περισσότερες τέτοιες συγκεκριμένες αλλαγές που είχαν ξεκινήσει από τη δεκαετία του 70. δείτε την ε, αναφορά των ε, διαφόρων συνιστοσών θα δείτε ότι υπάρχουν κλιματικές παράμετροι, επίσης όμως και υπεραλίευση οπωσδήποτε. Και για τις ε, κλιματικές και άλλες τέτοιες αλλαγές ως αίτια που μπορούν να συνεισφέρουν. Μια άλλη, ένα άλλο αίτιο είναι φυσικά η υπεραλίευση. Το πώς αλλάζει ο τρόπος αλίας και η ένταση αλίας που αλλάζει, οδηγεί στις αλλαγές οικοσυστημάτων στη συνέχεια. Και βλέπουμε ως ε, ε, σκηνικό ότι αυτά απαιτούνται για να κατανοήσουμε πώς ρυθμίζονται τα οικοσυστήματα εκ των κάτω προς τα άνω συνήθως. Και για τον, τη διαχείριση και έλεγχο των πόρων έχουμε και τη βιομάζα και όσον αφορά και την τροφική αλυσίδα και την διαθεσιμότητα στο κάτω άκρο της ε, τροφικής αλυσίδας για τη διαθεσιμότητα πόρων και επάνω επάνω βλέπουμε την ε, κορυφή, ε, έχουμε δηλαδή bottom top προσέγγιση και η αλληλεία αφορά τους στόχους, σκοπούς αλληλείας όσον αφορά μεγάλους όγκους αλλιευμάτων που αφαιρούνται από τα οικοσυστήματα και αυτό πάλι μπορεί να αλλάξει την δομή αυτών των οικοσυστημάτων. Και υπάρχει μείωση, συρρήκνωση των, ε, της τροφής που είναι διαθέσιμη πλέον από πλευράς ε, αυτών των αλλιευμάτων. Περισσότερες λεπτομέρειες ε, και επ' αυτού στη συνέχεια. Και έχουμε αλλαγές όσον αφορά και τη διαχείριση. Έχουμε λοιπόν και τον εκ των άνω προς τα κάτω έλεγχο αντί προς ε, εκ των κάτω προς τα άνω όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών. Έχουμε λοιπόν τα οικοσυστήματα, το πιο κοινό παράδειγμα είναι ε, σε σχέση με την ε, Βαλτική και την Μαύρη Θάλασσα που θα σας δώσω και λεπτομέρειες στη συνέχεια για την, την υφαλοκρηπίδα όσον αφορά την Σκοτία θα δείτε το τι συμβαίνει εκεί. Έχουμε παρουσία ε, πολλών ε, ηχθείων που ασχολούνται ακριβώς με την, ε, τη θύρα άλλων αλλιευμάτων. Έχουμε και τις αλλαγές όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές, επιπτώσεις της αλλίευσης, διακοιμάνσεις όσον αφορά την, τον πληθυσμό των νυχθείων, Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε σχέση με αυτά τα σημαντικά στοιχεία. Μια ιδέα αυτών των ε, στοιχείων που έχουν ε, αλληλένδετες επιπτώσεις και με αυτόν τον τρόπο εξετάζουμε την αθεκτικότητα και τις ε, μεταβολές όσον αφορά τα καθεστώτα οικοσυστημάτων. Υπάρχει εδώ και το θέμα της αντιμετώπισης των πιέσεων που μπορεί να καταδείξει την ανθεκτικότητα κάποιων πληθυσμών. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το ότι έχουμε ανθεκτικά ή υγιή οικοσυστήματα. Αυτό τι σημαίνει. Αν υποστούν πιέσεις όπως με τα μαύρα βέλη λόγω κλιματικών αλλαγών ή συνθήκων ή λόγω ε, βλέπετε ότι το οικοσύστημα αυτό δεν θα υποστεί μάλλον μεγάλες αλλαγές λόγω του ότι είναι ανθεκτικό και υγιές. Και στη συνέχεια βλέπουμε ότι όσον αφορά άλλα αίτια, ε, εξωτερικά αίτια, όπως ε, για παράδειγμα την αλία, την ε, υπεραλίευση, βλέπουμε ότι είναι πολύ εύκολο μέσω η μεγάλης έντασης να αλλάξει το οικοσύστημα, να υποστεί αλλαγές. Μπορεί να συμβεί αυτό καμιά φορά και από κλιματικές ε, ε, συνέπειες. Όσο, ωστόσο, οι εξωγενείς συνθήκες όπως η υπεραλίευση μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες αλλαγές. Σε σχέση με το feedback που υφίσταται, έχουμε εδώ τα πιο σημαντικά feedback ως ε, στοιχεία. Βλέπουμε και την μείωση λόγω της αλίευσης και των κλιματικών συνθήκων και υποθέτουμε, υπάρχει υπόθεση εργασίας ε, ότι ε, καθώς ε, ψάρια θηρευτές καταστρέφουν τον γόνο των ηχθείων που πολλαπλασιάζονται στην περιοχή όπου κυνηγούν υπάρχει συρρήκνωση του ηχθειακού όγκου. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα από τη μελέτη αυτό. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω κάποια πράγματα ως ε, προειδοποίηση για την διαχείριση. Αυτό που χρειάζεται συχνότερα για την εποπτεία, την επόπτευση και τη διαχείριση μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επειδή υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε συγκεκριμένες περιόδους, καμιά φορά αλλάζουν τα στατιστικά χαρακτηριστικά στοιχεία μπροστά σε μια επικείμενη αλλαγή και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έγκαιρη προειδοποίηση για μας να συναγάγουμε τα συμπεράσματα της επικείμενης ε, αλλαγής καθεστώτος οικοσυστημάτων και να ληφθούν προληπτικώς μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των αιτίων και κινδύνων. Συνοψίζω, κατά τη διάρκεια ε, ε, των αλλαγών αυτών που βλέπουμε που ξεκίνησαν μέσα στη δεκαετία του 80, αρχές της δεκαετίας του 90, βλέπουμε ότι αυτά τα Αυτές οι παράμετροι που αφορούν τα οικοσυστήματα αφορούν και την υπεραλίευση Υπάρχουν εξωγενείς, ε, πολυσχηδείς ε, τέτοιοι ε, εξωγενείς παράγοντες που απαιτούνται για να υπάρξει μια τέτοια μεγάλη αλλαγή. Αυτά όλα μπορούν να υπονομεύσουν την ανθεκτικότητα και τον υγιή χαρακτήρα οικοσυστημάτων και να οδηγήσουν σε κατάρρευση. Είναι σημαντικό να εξεταστεί ότι αυτές οι αλλαγές καθεστώτων είναι πολύ δύσκολο να αναστραφούν εφόσον έχουν ξεκινήσει. Και έχουμε και παραδείγματα ε, ότι ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη διαχείριση και στη στρατηγική που θα υιοθετηθεί για την στρατηγική και πρέπει να έχουμε μια δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης. Ευχαριστώ. Πρόεδρο σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια από πλευράς Κασίνη από το Σουηδικό Ίδρυμα Ιδρολογικών ε, ε, Θαλάσσιων Ερευνών θα λάβετε τον λόγο παρακαλώ για 15 λεπτά. Καλημέρα σας. Θα σας δώσω μια εισαγωγή όσον αφορά την αλλαγή η έχει συμβεί στη Βαλτική θάλασσα. Αυτό το οποίο θα εξετάσω αυτή τη στιγμή είναι το κεντρικό μέρος της Βαλτική Θάλασσας, διότι εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και εκεί έχουμε μόνιμη πληροφόρηση όσον αφορά την αλίευση, την απασχόληση και ούτω καθεξής του οικοσυστήματος. Και αυτή η περιοχή λοιπόν έχει αλλάξει πάρα πολύ και τελευταίο διάστημα και έχει αλλάξει κατά τρεις τρόπους, είναι το κλίμα, η εισαγωγή καθώς επίσης και η ελίευση. Εάν προσπαθήσουμε να δούμε αυτή τη στιγμή τις εξωτερικούς παράγοντες που έχουν αλλάξει, είναι, έχει πέσει το αλμυρό της θάλασσας, καθώς επίσης αυξάνεται τώρα, τουλάχιστον στα χαμηλότερα επίπεδα, αντιθέτως έχει αυξηθεί η θερμοκρασία της θαλάσσης στο επίπεδο, στο ψηλότερο επίπεδο της επιφανίας. Και εάν δείτε πραγματικά αυτά τα στιγμήματα τα όσον αφορά από το 80 μέχρι σήμερα όσον αφορά τον ευτροφισμό έχουν αυξηθεί λόγω της πολιτικών πολιτικών από τις διάφορες χώρες οι οποίες έχουν ακολουθήσει σε αυτές τις χώρες. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, οι τροφές αυτή τη στιγμή δεν έχει. Έτσι λοιπόν το ο φόσφορος αυξάνεται όλο και περισσότερο καθώς επίσης και το θείο μειώνεται. Και βεβαίως αυτά όλα καταλαβαίνουμε τη σημεία. Ένα άλλο μεγάλο σημείο είναι είναι περιοχές ακύρωση οι οποίες δεν έχουν αρκετό οξυγόνο και βλέπετε από αυτά τα μαύρα σημεία ποια είναι η έκταση αυτής της περιοχής. Αυτές τα τελευταία 15, 15 χρόνια έχει αυξηθεί. Υπάρχουν λοιπόν περιοχές που δεν έχουν καθόλου οξυγόνο ή πολύ λίγο οξυγόνο και βλέπουμε τις επιπτώσεις. Εάν δείτε λοιπόν τις, την, το εμπόριο όσον αφορά αυτόν, τον βλέπουμε ότι υπάρχει η ρέγγα η οποία είχε πνευθεί πάρα πολύ το 1980 και τα τελευταία δύο-τρία χρόνια άρχισε εκ νέου να δείχνει μερικά σήματα αύξησης. Η Σαρδελόρεγγα από την άλλη μεριά βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα. Επίσης τα αποθέματα αυξάνονται σε αυτά τα χρόνια τα οποία αυξήθηκαν. Εάν δείτε τους λόγους για τους οποίους αυτή η όλα αυτά, βλέπετε ότι για τον Ρέγκα, για το Κάδο, ήταν πολύ ψηλότερο από το επίπεδο το οποίο είχε προταθεί λόγω της θεσιμότητας που είχε και ο οργανισμός ο FBI υπάρχει μια προσπάθεια για την πρόληψη αυτής της θυμότητας των ψαριών και βλέπετε ότι στα τελευταία 20 χρόνια έγιναν πολλά πράγματα σε αυτό το τομέα. Το γεγονό ότι αυτή η επίπτωση όλων αυτών τα τελευταία τρία χρόνια έχουν δοθεί τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής ακολουθώντας λοιπόν το σχέδιο διαχείρισης της ΕΕ επέτρεψε το αποθέματα να αυξηθούν τα τελευταία τρία χρόνια. Επίσης, αυτό πλήττεται επίσης και από το κλίμα. Υπάρχει λοιπόν Ε, για να υπάρξει περισσότερη θα πρέπει να υπάρχει ε, ο σωστή οξυγόνης καθώς επίσης και το σωστό ποσοστό άλατος και αυτό έχει επίπτωση βεβαίω σε όλο τον κύκλο, στο πλακτόν και αυτό μπορεί βεβαίως μακροχρόνια να δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Βλέπουμε λοιπόν τα τελευταία 20 χρόνια την αύξηση του κάδου, κόδου, κάδου. Γιατί η αύξηση της, α, της θερμοκρασίας είχε επίπτωση και στα πρώτα και στα δεύτερα από αυτά τα είδη των ψαριών. Εάν πούμε πραγματικά από την άλλη μεριά τη μείωση της βιομάζας, έτσι όπως συνθέεται αυτή με τη θυσιμότητα των ψαριών, πράγμα το οποίο για πολλά χρόνια ήταν πολύ ψηλότερα από το επίπεδο από το οποίο προτιθνόταν από την αντίστοιχη επιτροπή και αν δούμε πραγματικά πώς οφείλεται αυτό στην αύξηση της, του ταλμυρότητας καθώς επίσης και της αλίευσης. Εάν δείτε πραγματικά ποια είναι τα γεγονότα αυτά της αλλαγή από το υψηλότερο στο χαμηλότερο θα δείτε ότι όπως είπε ο προλαλής ότι η έλλειψη αυτή του κάδου στα δεκαετία του 90 σήμαινε ότι και το πλακτόν έχει μειωθεί και βεβαίως αυτά υπήρξαν παράλληλα και υπήρξε μια αύξηση του φυτόπλακτών. Αυτό είναι λοιπόν ένα από τα πράγματα τα οποία προσπαθεί να προκληθεί ε, αυτή η πτώση του όλου οικοσυστήματος. Όλη αυτή λοιπόν η τροφική αλυσίδα θα πρέπει να δούμε ότι τι γίνεται με την ε, και τη ραγιά. Υπάρχει πραγματικά μια, ένας ανταγωνισμός μεταξύ των δύο αυτών και, και οι δύο αυτά ήδη έχουν μειωθεί και σήμερα βρισκόμαστε και τα δύο αυτά ψάρια είναι και μικρότερα σε μέγεθο, αλλά και πολύ πιο αδύναμα και αδύνατα. Εάν δίνατε λοιπόν τι αλλαγέ, τι δομέ που έχουν γίνει όσον αφορά αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν η αλμυρότητα του θαλάσσια ήταν πολύ ψηλά και η, ο κάδος ήταν πολύ χαμηλός. Και αυτό βεβαίως κάτσε και στη Σαρδελόραγκα πολύ πιο χαμηλά έτσι λοιπόν η βιομάζα καθώς και το φυτοπλακτόν ήταν επίσης πολύ χαμηλά λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας. Αλλά σε πρόσφατα, μετά τη δεκαετία του 1990, λόγω της αύξησης της θερμο... κλίματος, της θερμοκρασίας, υπήρξε μια αύξηση και στρατητήθηκε σε χαμηλό επίπεδο η βιομάζα του φυτοπλακτών, καθώς καθώς επίσης και υπάρχει, υπήρχε μία μείωση του ρήτου σε αυτή την περιοχή. Τι σημαίνει αυτό για το σύστημα και για τα άλλα συστήματα, ότι μπορεί να υπάρξουν επιπτώσεις, δηλαδή Αυτή η κατάσταση πολύ δύσκολη να επιστροφεί, διότι υπάρχει ένας μηχανισμός επιπτώσεως, ο οποίος πραγματικά διατηρεί αυτή την κατάσταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν όπως βλέπουμε σημαίνει πως εάν οι συνθήκε είναι πολύ καλά μπορεί εκ νέου να αυξηθεί η βιομάζα του φύλλου στο πλακτόν, πράγμα το οποίο θα έχει θετική επίπτωση στο όλο κύκλο. Αλλά όταν πέσει ο κάδος, η πρακτική αυτή και αν έχουμε πολύ καλές συνθήκες, το πλακτόν δεν μπορεί να αυξηθεί και αυτό έχει ε, επειδή η σαρδελόρακα δεν μπορεί να αυξηθεί και αυτό σε έχει αισθητοτά επίπτωση στα άλλα ψάρια όπως είναι ο κάδος και η ρέγγα. Όλοι αυτοί οι τρίπτες μηχανισμοί λοιπόν προσπαθούν να διατηρήσουν ούτως ώστε η σαρδελόρακα να μένει σε μία προτεραιότητα για να μπορεί να σε όλο σύστημα. Αυτό ο μηχανισμό λοιπόν τον οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά βιολογικά στοιχεία τα οποία η αύξηση των, της βιομάζας ή το οξυγόνο, η θερμοκρασία και όλα αυτά τα στιγμή βλέπετε είναι πολύ το πρόβλημα αλλά όλα αυτά μπορούν να αυξηθούν και ιδιαίτερα σύνθετο προβλημα αλλα ολα αυτα μπορουν υπάρχει μια βελτίωση μετά τη δεκαετία του 90 λόγω του κλίματος και αυτό νομίζω πως πραγματικά είναι ένας δείκτης για την βελτίωση όλης αυτής της καταστάσεως. Άλλες επιπτώσεις υπάρχουν ε, σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο, δηλαδή σημαίνει πως με την αύξηση των στοιχείων εκείνων τα οποία είναι διατροφικά στοιχεία μέσω της ανθρώπινης κατανάλωσης, αυτό λοιπόν αυξάνει πολύ το φυτοπλακτόν και, και αυτές είναι πολύ οξικές, ε, τοξικές κατατάξεις και αυτό ε, δημιουργεί μία αναστολή του, του φωσφόρου. Και εάν ακόμη μπορούμε να τα διατηρήσουμε αυτά και μπορούμε να χαμηλώσουμε αυτές τις ε, εκπομπές των ανθρωπίνων αποβλήτων. Εν μία άλλη επίπτωση θα μπορούν να ήταν να διατηρήσει τον φύλλο του πλακτών, του με, σε περιοχές που υπάρχει λίγο οξυγόνο βεβαίως βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ λιγότερα ψάρια και ιδιαίτερα ο κάδος. Έτσι λοιπόν εφόσον αυτό συνδέεται βεβαίως και με την αύξηση των φυτοπλανκτών λόγω έλλειψης του οξυγόνου. Βλέπετε λοιπόν ότι στα τελευταία 40 χρόνια έχει υποστεί μεγάλη αλλαγή στην Βαλτική θάλασσα οφείλονται όλα αυτά στην, στην μάλλον, η οποία, το οποίο έχει σχέση με την, την αλυσίδα και την κλίμακα. και βλέπουμε αυτή τη στιγμή και τη λειτουργία του όλου οικοσυστήματος ό,τι έχει αλλάξει Προσπαθούμε λοιπόν να διατηρήσουμε ε, ε, είναι δύσκολο. Αυτό το σύστημα διατηρηθεί και είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουμε στο παλαιότερο σύστημα, να το ανατρέψουμε αν θέλετε. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει όμως αυτή τη στιγμή, να παραμείνει πάρα πολύ χαμηλή η αλίευση ως αφορά τον κάδο και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόγραμμα διαχείρισης της ΕΕ το οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί διότι τα δύο-τρία τελευταία χρόνια όσον αφορά τον κάδο τον και υπάρχει μια πίεση σε αυτή την περιοχή για την ανάκαμψη και ένα κάτι άλλο θέμα είναι να προσπαθήσει να εισαχθεί να γίνει μια προσαρμογή ε, μια προσαρμογή η οποία θα έχει θα απαλλάξει την σημότητα η οποία οφείλεται στην έλλειψη οξυγόνου, στη, στην αλάτωση του ύδατος και ούτω καθεξής. αυτή οι δύο παράγοντες σε δηλαδή, συνειρμό. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε, να ακολουθήσουμε αυτή τη, την προοπτική, μπορεί τα αποθέματα να αποκατασταθούν, όχι στα επίπεδα του 80 βεβαίω, αλλά σε κάποια ψηλά επίπεδα και μετά από αυτά τα συστήματα μπορούμε να αυξηθεί η ρέγγα, καθώς επίσης μπορεί να αυξηθεί και η σαρδελό ρέγγα και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ θα βοηθήσει πάρα πολύ και επίσης εφόσον υπάρξει μια λιγότερη δυνατότητα αποβολής και βεβαίως όλη αυτή η αλυσία θα καταντήσει στο κάδο. Θα τελειώντας θέλω να πω θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι ορισμένες εξωτερικές πτώσεις σε αυτό το οικοσύστημα, διότι σε αυτές τις περιοχές που δεν υπάρχει οξυγόνο, μπορεί να γίνει πραγματικά μια εισαγωγή από τη Βόρεια Θάλασσα, αλλά δεν είναι αρκετό, μπορεί απλώς να μειώσει τη θνησιμότητα αυτών των ψαριών, όταν βεβαίως το οξυγόνο είναι αρκετή στο επίπεδο του βυθού. Αυτό βεβαίω ε, μπορεί να βοηθήσει διότι υπάρχουν μερικές προβλέπεις οι οποίες βλέπουν ότι, ότι θα αυξηθεί και, το, και η θερμοκρασία και η αλμυρότητα της θάλασσας. Και αυτό βεβαίως θα είναι περιοδικό για τον κάδο καθώς επίσης και σε αρδελόραγγα. Εάν αυτά λοιπόν βελτιωθούν, βεβαίως όλα αυτά θα μπορούν να αλλάξουν το όλο οικοσύστημα στη Βαλτική θάλασσα, ωστόσο μπορούν να είναι ευεργετικά. Αυτά ήταν όλα όσα είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, δόκτωρα Καζίνη, για την παρουσίαση του οικοσυστήματος στην Βαλτική. Το λόγο έχει τώρα ο Γιώργη Δάσκαλοφ από την Ακαδημία Επιστημών της Βουλγαρίας. Έχει το λόγο για 15 λεπτά. thank everyone. My talk is about... Uh, Θα σας μιλήσω για τη μετατόπιση των οικοσυστημάτων στην ε, Μαύρη Θάλασσα. Στον Εύξηνο δηλαδή. μια περιγραφή της μετατόπισης του οικοσυστήματος και της τροφικής κλίμακος που του δημιουργεί στη Μαύρη Θάλασσα, στον Εύξηνο. Να πω λίγα λόγια σχετικά με το, τα αίτια, όπως τα παρατηρήσαμε στον Εύξηνο και να περιγράψω επίσης και κάποιες εναλλακτικέ συμπροματικές να δώσω εξηγήσει δηλαδή, για άλλους παράγοντες, όπως είναι Φερρυπίν, αν θέλετε τα εισβάλλοντα είδη, το κλίμα και η ευτροφισμός, θα μιλήσω επίσης για τη διαχείριση της αλληλείας και το πώς αυτό επηρεάζει τα συστήματα που υπόγειται δηλαδή σε αυτή τη μετατόπιση και θα δώσω και κάποιες συστάσεις. Αυτές, αυτά τα regime shifts και τα tropic cascades όπως περιγράφονται στη Μαύρη Θάλασσα, στον Εύξηνο δηλαδή, που ήταν το πρώτο μεγάλο θαλάσσιο οικοσύστημα που διαπιστώθηκαν για φαινόμενα και περιεγράφησαν επίσης, και πρέπει να λάβουμε υπόψη μα δύο μεγάλε μετατοπίσει shift στην ε, Μαύρη Θάλασσα. Η πρώτη συνέβη κατά τη δεκαετία τη δεκαετία του 1970, όπου οι πιο σημαντικοί αν θέλετε θηρευτέ και τα θαλάσσια θηλαστικά δηλαδή και οι μεγάλοι θηρευτέ δηλαδή κατεστράφησαν λόγω τη υπεραλίευση και αυτό δημιούργησε αυτό το τρόφι cascade για τα μικρά βασίλεια ήδη, αύξηση του ζωοπλανκτών και αύξηση επίσης και του φυτοπλανκτών και αλλαγές επίσης αν θέλετε στο περιβάλλον, αν θέλετε Αργότερα, αυτό το Trophic Cascade, η υπόθεση μάλλον, επιβεβαιώθηκε από ανάλογες αλλαγές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 που είχαμε και εκεί υπεραλίευση και αυτό δημιούργησε τις συνθήκες για την ανάπτυξη ζελατινόδους αν θέλετε πλανκτών που οδήγησε σε περαιτέρω υποβάθμιση αν θέλετε του ζωοπλανκτών, αύξηση του φυτοπλανκτών και αλλαγές επίσης και στην χημεία των υδάτων. Οι αλλαγές αυτές οδήγησαν και προκάλεσαν οι αλλαγέ αν θέλετε στο πάνω μέρο του συστήματος είχαν συνέπειες στη δομή των οικοσυστημάτων, στη λειτουργία τους, την ε, βάση της παραγωγής και την ποιότητα επίση των υδάτων. Όπως τα είδατε από τις προηγούμενες ομιλίες, τα φαινόμενα αυτά είναι αρκετά περίπλοκα. και λόγω αν θέλετε της πολυπλοκότητας των οικοσυστημάτων. Να δώσω θα ήθελα τώρα κάποιες λεπτομέρειες, κάποιες εξηγήσεις αναφορικά με το μηχανισμό που δημιουργεί αυτά τα regime shift στην Μαύρη Θάλασσα. Πρώτα απ' όλα, οι αλλαγές αυτές είναι συστημικές αλλαγές. Στην δομή δηλαδή και στη λειτουργία των συστημάτων και κατευθύνονται εκ των άνω, εκ των άνω προς τα κάτω. Πρόκειται δηλαδή για αλλαγές οι οποίες συνεπάγονται διαφορετικά επίπεδα τροφισμού και το χαρακτηριστικό για την μετατόπιση του οικοσυστήματος είναι ότι αυτό οφείλεται στη θετική ανάδραση η οποία αν θέλετε διεύρυνε και ε, ύφτισε την αρχική πίεση. Παρατηρήσαμε επίσης και μια μη γραμμικότητα των μορφών που λαμβάνει αυτή, αυτό το regime shift. Τα πράγματα τα οποία φύγεται αν θέλετε σε κάποια χρονικά κενά που οδηγούν σε αυτή την υστέρηση. Και ένα από τα αίτια αυτών των time lags θα μπορούσε να είναι η ανθεκτικότητα του συστήματος. Το σύστημα είναι ανθεκτικό, ελαστικό δηλαδή. Και οι συνέπειε, αν θέλετε, ακολουθούν, να θέλετε, τα αίτια μετά από την παρέλευση ενό κάποιου χρονικού διαστήματο. Όπω έλεγα λοιπόν στην ε, Μαύρη Θάλασσα, ο βασικό μηχανισμό που παρατηρήσαμε είναι η αλίευση, αν θέλετε και αυτό το, η συνέπεια και η επίπτωση σε τον άνω προς τα κάτω, το top-down δηλαδή, αλλά τα συστήματα αυτά έχουν πολλαπλούς, πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν θέλετε, τη συμπεριφορά τους. Και οι παράγοντες αυτοί ενεργούν, αν θέλετε, με τρόπο αν θέλετε, που δημιουργεί αν θέλετε, πολλαπλά αποτελέσματα και οδηγεί σε πολλαπλά αποτελέσματα, αλλά τελικώ είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Το κλίμα, ο αυτοφισμός, κλιματικές αλλαγές και στην περίπτωση της Μάρης Θάλασσας, αν θέλετε, τα εισβάλλοντα είδη, συμμετέχουν και συμβάλλουν σε αυτές τις μετατοπίσεις, σε αυτά τα shifts και συμβάλλουν λίγο ή πολύ στην ανάπτυξη εναλλακτικών καθεστώτων. Αυτό που βλέπουμε από τα δεδομένα, ο πρώτος από τους παράγοντες είναι το κλίμα. Πρώτα απ' όλα η Μαύρη Θάλασσα είναι κάπως απομονωμένη. Είναι η μια ημί και κλεισμένη θάλασσα, η και κλεισμένη θάλασσα, αλλά αυτό επηρεάζεται νομίζω από το κλίμα του Ατλαντικού. Βρήκαμε έναν καλό συσχετισμό μεταξύ του κλίματος του Ατλαντικού Βόρειος Ατλαντικός και Δυτική Ρωσία, όπως βλέπετε στον πίνακα, στη διαφάνεια, πάση και αυτή η κλιματική αλλαγή επηρεάζει το τοπικό υδροκλίμα, δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα κάτω τη θερμοκρασία της θάλασσας δηλαδή και των ποταμιών και συσχετίζεται με την ε, αύξηση των αποθεμάτων των ε, ψαριών. Επίσης το κλίμα και το πώς επηρεάζει αυτό και αλληλεπιδρά με την αλία. Βλέπουμε στην περίοδο κατά την οποία η αυτονία των ψαριών επηρεάζεται από το κλίμα, έχουμε και τη μεγαλύτερη ηλιαυτική πίεση και τη μεγαλύτερη θνησιμότητα. Και αυτό βεβαίω οφείλεται στο γεγονός ότι μειώνεται το απόθεμα για κάποιους φυσικούς λόγους και για φυσικά αίτια, αλλά η αλληλεία δεν είναι προσαρμοσμένη σε αυτή την τροχιά, σε αυτή τη διαδρομή λειτουργεί συντηρητικά και κάποια στιγμή επηρεάζει αυτό τα, τα φθήνοντα ε, τα αποθέματα, τα μειούμενα αποθέματα και έχουμε κατάρρευση των αποθεμάτων και τη αλεία βεβαίω κάποια στιγμή. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια τη δεκαετία του 90, όπω είδατε στην προηγούμενη ομιλία. Τέλη τη δεκαετία του 80, αρχέ τη δεκαετία του 90, αυτέ οι μετατοπίσει εμφανίστηκαν σε πολλά τέτοια συστήματα παγκοσμίω. Ε, μια άλλη κατευθυντήρια δύναμης η οποία έχει περιγραφεί είναι ο ευτροφισμός. Στο σύστημα αυτό ο ευτροφισμός η επίδραση του ευτροφισμού στο σύστημα δηλαδή δεν αφορά τόσο πολύ την δομή αλλά ολόκληρο το σύστημα το επηρεάζει. Και ειδικότερα όταν το σύστημα αυτό δεν έχει αν θέλετε αυτούς τους μεγάλους θηρευτές, στην περίπτωση αυτή έχουμε άφθονο φυτοπλανκτών και τον πληθυσμό αν θέλετε από μέδουσε jellyfish. Και αυτό βεβαίω επηρεάζει και τους δύο αυτούς, ε, τις δύο αυτές ακόμη περισσότερο. Και αυτό βεβαίω θα μπορούσε να ενισχύσει, να θέλετε, τη σωτική ανάδραση στο σύστημα, να δημιουργήσει περισσότερη υποξία και αυτές τις αρνητικές συνέπειες στο θαλάσσιο περιβάλλον, στο υδάτινο περιβάλλον. Σε κάποια πρόσφατα μοντέλα τα οποία μελετήσαμε, διαπιστώσαμε, είδαμε ότι αν προσθεθεί ένα top level άφθονο στο σύστημα, τότε νομίζουμε θα μπορούσε να στηρίξει. Σε κάτω συνθήκε όμω υψηλότερου μεγαλύτερου στροφισμού. Μια άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση στη Μαύρη Θάλασσα ήταν η εισβολή αυτών των ειδών, αν θέλετε, μεδουσών, μειόψης lady, δηλαδή κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, ο μηχανισμός αυτός σχετίζεται και πάλι με την αλία και την υπεραλίευση και μπορούμε να παρατηρήσουμε την μείωση των αποθεμάτων των ηχθείων λόγω της υπεραλίευσης και άλλων παραγόντων όπως είπα προηγουμένως, αύξηση της θρησιμότητας επίσης των ηχθείων και έχουμε και με τη μαζική αυτή εξέλιξη του πληθυσμού αυτού του εισβάλλοντος είδους αυτής της μέδουσα δηλαδή και το ίδιο συνέβη και στην ε, Κασπία και τώρα και τη Βόρεια Θάλασσα και τη Θάλασσα της Βαλτικής και έχουμε και ένα άλλο είδος μέδουσα επίσης ένα αλόχθονο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 εμφανίστηκε αυτό εξειδικευμένο θηρευτή. Βλέπετε ότι η φύση, αν θέλετε, προσπαθεί να ρυθμίσει την κατάσταση αυτή και να λύσει τα προβλήματά τη. Και υπάρχει έλεγχο αυτού του πληθυσμού. διότι παρουσιαστήκε αν θέλετε και μια ανάκαμψη των αποθεμάτων των μικρών βαθιδίων. Τώρα αυτές οι μετατοπίσεις των καθεστώτων ε, είναι σημαντική, αποτελούν σημαντική πρόκληση, διότι τα συστήματα αυτά, όπως βλέπετε, είναι ιδιαίτερα περίπλοκα, λίαν περίπλοκα. Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί τους οποίους ακόμη δεν γνωρίζουμε, αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η αλία είναι ένας παράγων. Όχι μόνο τα αποθέματα, αλλά ολοκλήρου του οικοσυστήματος θα μπορούσε να μετατοπίσει το σύστημα αυτό σε ανεπιθύμητες καταστάσεις. Αλλά υπάρχει όμως και κανονισμός και διαχείριση για την αλία. Υπάρχουν πάμπολα παραδείγματα επιτυχιών και αποτυχιών σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της αλίας, αλλά είναι πιθανό και δυνατόν να γίνουν όλα αυτά. Άρα, αυτό που χρειαζόμαστε πρώτα απ' όλα είναι να καταλάβουμε καλύτερα αυτές τις μετατοπίσεις καθεστώτων, τα regime shifts, θα πρέπει να τα μελετήσουμε και κατόπιν και ενδεχομένως θα μπορούσαμε να προβλέψουμε μέχρι ενό βασμού ε, όταν θα συμβαίνουν δηλαδή όπως είχαμε αυτό την εργασία που έγινε για τους δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης και νομίζω ότι θα μπορούσαν πολλά ακόμη να αναπτυχθούν στο μέλλον, θα γνωρίζουμε καλύτερα και τους μηχανισμούς. Η διαχείριση θα πρέπει βεβαίω να είναι προσαρμοσμένη, θα πρέπει να προσαρμόσουν τη διαχείριση σε μακροπρόθεσμα καθεστώτα και ένα απλό τρόπο για να το περιγράψει αυτό κανεί. δεν ξέρω πώ θα συμβεί αυτό στην πράξη, είναι να αναγκάσουμε την αλληλεία να μειώσουμε την, αλλαγή, αλλιευτική πίεση, κατά τη διάρκεια θέλετε, καθεστώτος να θέλετε χαμηλής παραγωγικότητος και να διατηρήσουμε δηλαδή στην κατάσταση του Στάτου βο ή και σε μια αύξηση να έχουμε ένα παραγωγικό καθεστώς. Νομίζω πάντως ότι τελικός στόχος της διαχείρισης είναι να ανατραπεί, να ανακτηθούν τα οικοσυστήματα και να φτάσουμε, αν θέλετε, τα αποθέματα, των αποθέματα σε αποδεκτά επίπεδα. Βιώσιμες δηλαδή αποδόσεις να έχουμε και καλά επίπεδα αποθεμάτων. Η εμπειρία μας πάντως στην Μαύρη Θάλασσα έδειξε ότι οι αλλαγές οι διαστοτικές αλλαγέ στα οικοσυστήματα δεν θα οδηγήσουν ακριβώς στην προηγούμενη κατάσταση, αλλά είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες. Αλλά τα συστήματα αυτά έχουν μνήμη, θα θυμίζω. Τίνουν να φτάσουν στο προηγούμενο επίπεδο και καλύτερο πολλές φορές επίπεδο, αλλά τα εισβάλλοντα ήδη, και άλλα φαινόμενα μπορούν ή και το κλίμα επίση να διατηρήσει αν θέλετε το καθεστώ σε ανεπιθύμητα επίπεδα, δηλαδή για ένα κάποιο χρονικό διάστημα. Τα συμπεράσματά μας τώρα. Η υπεραλίευση. Έχουν διαβρώσει το οικοσύστημα της ε, Μαύρης Θάλασσας δημιούργησαν ανθυγιεινές περιβαλλοντικές καταστάσεις και κοινωνικές επίση με την κατάρρευση της αλίας. Έβλαψαν επίσης την ποικιλότητα και θα πρέπει τα ανθεκτικά συστήματα να αποκαταστήσουν όλα τα συστατικά τους, να μειωθεί η ανθρωπογενής επίπτωση, η ελεπίδραση των αποθεμάτων, να αυξηθεί η διαφοροποίηση και η περιβαλλοντική ποιότητα να, και βεβαίω αυτό θα χρειαστεί η επιστήμη δηλαδή να μπορεί να προσαρμοστεί στις ε, μεταβαλλόμενες συνθήκες και να αντιμετωπίσει το μεταβαλλόμενο βαθμό πολυπλοκότητος του συστήματος. Δηλαδή για να μπορέσουμε να ολοποιήσουμε και να εφαρμόσουμε ένα επιτυχές σύστημα θα είναι πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δυσχερές, γιατί η κατάσταση των αποθεμάτων και το θαλάσσιο περιβάλλον είναι τέτοια σημασία που αυτέ οι προκλήσει θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από εμά, από την κοινωνία δηλαδή στο σύνολό τη. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Eh, Ευχαριστούμε, Δόκτωρ Δασκάλοφ. Ε, το λόγο έχει τώρα ο κύριο Μπρίτα Έριξον από το Πανεπιστήμιο Γκρόνιγκεν των Κατοχωρών σχετικά με το ζήτημα της περαλήψης και των ε, φυγιών. So good morning. Καλημέρα σα. Θέλω να σα πω περί πώ αυξάνεται και αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή όλο περισσότερο τα φύκια. Η μου μίλησε για την αλλαγή, ποια υπάρχουν στοιχεία, ποια δεδομένα και έχουν αλλάξει. Αυτή τη στιγμή αυτή έχετε μια ε, αύξηση έχετε μια αύξηση των ψαριών τα οποία είναι κρεοφάγα και μια μείωση αυτών που είναι φυτοφάγα. Ποια είναι η φύση λοιπόν αυτή τη στιγμή. Ο, αυτά όλα που θα αποτελούν την αύξηση των φυκιών. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή να δούμε και θα σα παρουσιάσω τα αποτελέσματα αυτή τη έκθεσης και ποια είναι οι αρνητικέ επιπτώσει όλων αυτών των προσπαθειών που έχουν και Όλη αυτή η αλλιεύση βοηθάει στην αύξηση των φυκιών και όλα αυτά έχουν μια συνέργεια μεταξύ τους, συνεργάζονται για αυτή την ανάπτυξη, την υπερβολική ανάπτυξη των φυκιών. Έτσι, μπορούμε να πούμε τι σημαίνει αυτή η υπερανάπτυξη των φυκιών. είναι ότι στο όλο οικοσύστημα υπάρχουν πάρα πολλά φυκιά τα οποία δεν υπήρχαν παλαιότερα και αυτό δημιουργεί προβλήματα και αυτά τα προβλήματα είναι ε, επιβλαβή. Αυτό. Αυτό κοστίζει περίπου 665 εκατομμύρια και αυτό είναι βεβαίως μια εκτίμηση που γίνεται του κόστου της τη Πρόκειται για μικροσκοπικούς οργανισμούς, για μονοκύτταρους οργανισμούς που αναπτύσσονται. Είναι η Timeton Flagellates, άλλα άλλα βακτήρια και αυτό περισσότερο από τα φυλαμέντου σάλτσια, αυτά τα φυκιά. Θα σας δείξω ακριβώς τι λέγω. μπράβο. Υπάρχουν λοιπόν μερικές φύκια τα οποία παράγουν τοξίνες. Υπάρχουν είναι αυτές οι τοξίνες οι οποίες εισάγονται μέσα σε αυτή την τροφική αλυσία και βεβαίως περνάνε από τα ψάρια στους ανθρώπους και δημιουργούν προβλήματα τα οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Επίσης υπάρχουν άλλα τα οποία σκοτώνουν τα ψάρια και τους οργανισμούς οι οποίοι άπτονται Και αυτό αποτελεί πρόβλημα για την υδατοκαλλιέργεια. Μπορεί να έχουμε και αυτά τα είδη των φυκιών που είναι υψηλής πυκνότητος, αλλά βλέπουμε εδώ την Σουηδία, Βαλτική θάλασσα και όλο το πράσινο εδώ είναι ένα μεγάλο, θέλετε, κομμάτι, αν θέλετε, βακτηριδίων. Βλέπετε και τη Φιλανδία και την Ιστονία. Βλέπουμε τεράστιες ποσότητες οργανικού υλικού που είναι συσσωρευμένο. Και τι συμβαίνει όταν έχουμε τέτοια υπερβολική παραγωγή, αν θέλετε, φυκιών. Θα μπορούσαμε να έχουμε πολλά προβλήματα. Καταρχήν ε, υπάρχει ανάγκη αποσύνθεσης αυτών. Θα πρέπει κάποια στιγμή να εξαφανιστούν και χρησιμοποιούν το οξυγόνο που βρίσκουν στο νερό. Και έχουμε αυτές τις συνθήκες της ανοξίας, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ επιζήνιο για όλους άλλους οργανισμούς. Στις κάτω χώρες, δηλαδή το 2001, είχαμε μια θνησιμότητα 10 εκατομμυρίων, αν θέλετε, μυδιών δηλαδή, από ένα και μόνο τέτοιο είδος φύκη, το οποίο επηρεάζει την υδατοκαλλιέργεια και επηρέασε. Μπορεί να έχουμε και τη σχηματισμό επισμικήτων, δηλαδή χάνονται πολλοί οικότοποι, αν θέλετε, που έχουμε επίσης και προβλήματα τα οποία αν θέλετε μπερδεύουν θέλετε, το αλλιευτικό υλικό. Έχουμε δηλαδή την ε, παράλληλα του καγεράκια εδώ και βλέπετε όλο αυτό το ελαφρύ αν θέλετε κίτρινο νήμα εδώ πέρα κάτω που σημαίνει φύκια τα οποία αυξάνονται. Βλέπετε και ένα άλλο παράδειγμα εδώ για το σχηματισμό, αν θέλετε, Μικήτων από την θάλασσα του Μαρμαρά. Βλέπετε ότι ο σχηματισμός των Μικήτων ε, οφείλεται, θέλει, σε μια γελατίνη που δημιουργείται στο νερό μέσα. Έχουμε αυτό το γλιώδες, το υλικό, το κολλώδες υλικό. Και υπάρχει μεγάλη δυσκολία, αν θέλετε, να μπορέσει να σηκώσει, αν θέλετε, το αλληλευτικό, τα αλληλευτικά εργαλεία. Δεν μπορεί μάλιστα να τα, φέρεις, να τα σηκώσει μηχανικά, δηλαδή θα πρέπει να τα με το χέρι, δηλαδή, και διαφορετικά μπορεί να τα καταστρέψει. Και το 2007 και το 2008 οι αλληλείς έχασαν το μεγάλο ποσοστό, αν θέλετε, από τα κέρδη τους. Και εκτιμάται ότι αυτοί οι επιβλαβείς οργανισμοί θα δημιουργούν απόλυες για την αλληλεία 177 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Αυτό βεβαίω δεν περιλαμβάνει και δεν καλύπτει ούτε την Αδριατική αλλά ούτε και τη Μαύρη Θάλασσα. Επομένω, το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο αυτή η υπεραλίευση συμβάλλει στη δημιουργία και στην ανάπτυξη του προβλήματο αυτού. Προσπαθήσαμε να δούμε τι συνέπειε με διάφορα τα οποία έχουμε για να σας παρουσιάσουμε πάρα πολύ σύντομα αυτή την ανάλυση που έχει γίνει του δικτύου αν θέλετε. Είναι μια εκπροσώπηση ποιος κάνει τι σε σε αυτή την αλυσίδα. Το κάναμε αυτό βλέποντα όλα στοιχεία τα οποία με το ισχού που είχαμε από όλη την Ευρώπη. Θα δείτε λοιπόν στην σχέση που υπάρχει στη Βόρεια Θάλασσα για αυτά τα θέματα. 26 από 27 ομάδες θα μείωσε σε 7 και μπορούμε να δούμε ότι, ότι υπάρχουν τρεις ομάδες, υπάρχουν τα τοξικά φύκια, τα ημέδουσες και όλες αυτά τα οποία δημιουργούν αυτή η γραμμική αυτός ο γραμ, γραμμικός κύκλος αν θέλετε της διατροφής αυτό το οποίο συμβαίνει όταν εξετάσουμε αυτό το σύστημα είναι ότι εάν μειώσουμε αυτά τα αρπακτικά ε, ψάρια βλέπουμε ότι αυξάνονται τα φύκια και αυτό συμβαίνει αν ταυτόχρονα υπάρχει επίπτωση στο σύστημα ως εξής. Διότι υπάρχει μία αλλαγή η οποία γίνεται, αλλά δεν ακολουθεί όλη τη γραμμή, εάν εν ταυτό εάν αυτό το βλέπετε στην Περτική θάλασσα ιδιαίτερα Λόγω του ευτροχισμού βλέπετε ότι αυτό μειώνει το γάδο, αυξάνεται πολύ περισσότερο η ε, Και θυμηθείτε, η Βαλτική είναι μια περιοχή η οποία υπάρχει περισσότερο ευτροφισμός. Επίσης από τη Βόρεια Θάλα υπάρχουν δείκτες, διότι δεν είναι επεξεργαστεί βεβαίω αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα σημεία, αλλά μπορούμε ότι υπάρχει όλο από το 90 και μετά όλο μειώσει αλίευση του γάδου. Ενδιαφέρον λοιπόν, εάν δούμε πραγματικά αυτό το σύστημα, όλο και περισσότερο τα μικρά μειώνονται τα μικρά ψάρια όπως είναι η σαρδρόγαδος και η ατσούγα και αυτό που βλέπουμε ότι υπάρχει αυτοψινός και περισσότερη τοξικότητα και όλο και περισσότερες μέρουσες. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε αυτό το, το σύστημα να το εντάξουμε, πώς μπορούμε να βρούμε εκείνες τις συνιστώσεις και εφόσον αυτή τη στιγμή γύρω στο 90 είχε αυτό το σύστημα καταρρεύσει ολόκληρο, πώς μπορούμε να το ανατρέψουμε. Για να το πω λοιπόν ανακεφαλαιόντως έχω να πω τα εξή. Η ανάλυση η οποία θέλουμε να κάνουμε είναι ότι η έλλειψη των αρπακτικών ζώων, ε, ψαριών αυξάνει όλο και περισσότερο τα φύκια, σύμβολη θα και αυτό βεβαίως έχει επίπτωση. Βεβαίως είναι όλα αυτά στοιχεία τα οποία είναι περιορισμένα. Άρα θα πρέπει να δούμε τι γίνονται σε άλλες θάλασσες. Μπορούμε να το κάνουμε όμως στις ακτές και θα σας δείξω ένα παράδειγμα εδώ όπου Ε, πώς η υπερθύρευση στην ανοιχτή θάλασσα δημιουργεί τα φύκια στις παράκτης περιοχές. Αυτή είναι από την, ε, περιοχή 27. Βλέπετε αυτή τη στιγμή όλο και περισσότερο αυξάνεται το ένα ψάρι, μειώνεται το άλλο και υπάρχει μια, το sticker bank το οποίο είναι ένα άλλο μικρό ψάρι έχει αυξηθεί πάρα πολύ και είναι ενδιαφέρον διότι αυτό δείχνει ότι το χειμώνα είναι στην ανοιχτή θάλασσα και μένουν εκεί το χειμώνα, το, το καλοκαίρι έρχονται στην ακτή και αναπαράγονται. Και αυτό συμβαίνει στην παρτική. Είναι τα Tigerbags, είναι τόσο περίπου, 5, 6, 7 εκατοστά και βεβαίως αυτή η περιοχή όπως βλέπετε είναι γεμάτη φύκια. Τελικά όλα αυτά τα οποία βλέπετε εδώ είναι ενδιαφέρον αυτό που αποκαλύπτει είναι ότι υπάρχει μια διασύνδεση ότι η αύξηση αυτού του ψαριού αυξάνει και τα θήκια που σας ανέφερα προηγουμένως. Σε όλη τη Σουηδική Ακτή και στη Φιλανδία βλέπουμε αυτό το φαινόμενο να αναπτύσσεται και βλέπουμε ότι αυτό το stickleback το ψάρι όλο και περισσότερο κυριαρχεί καθώς επίσης και η αύξηση αυτού του φυκιού. Σε άλλες περιοχές που δεν έχουν το stickleback και που υπάρχουν τα αρπακτικά ψάρια υπάρχει μόνο ένα 10% αύξηση των φυκιών. Αυτό είναι δείγμα ότι υπάρχει μια αλληλοσύνδεση με το δύο. Εάν προσθέσετε περισσότερα αυτά τα μικρά ψάρια, όλο και περισσότερα αυξάνεται ή το φύγει στις παράκτητες περιοχές. Έχουμε λοιπόν ένα, μια βάση και δείχνουμε ότι αυτό το οποίο έχει γίνει μέχρι στιγμής είναι εάν πάρουμε όλα αυτά τα ψάρια από τη φύγη περιοχή και τα μικρά ψάρια και προσπαθούμε να εισάγουμε άλλα ψάρια εκεί, βλέπουμε ότι γίνεται, υπάρχει μια εξισορρόπηση. Έτσι, Βλέπετε εδώ, σε αυτό το σημείο υπάρχουν πάρα πολλά φύκια τα οποία έχουν αναπτυχθεί. Επίσης αυτή τη βάση έχουμε όταν βγάλαμε τα ψάρια από αυτή την περιοχή βλέπουμε ότι μειώθηκαν και τα φύκια. Το παραλαμβάνω αυτό και είναι... Βλέπουμε εδώ διάφορες περιπτώσεις που σας δείχνω αυτές όλες Εάν λοιπόν βλέπετε αφαιρέσετε τα αρπακτικά ψάρια, αυξάνονται τα μικρά ψάρια και αυξάνεται όπως είπα και τα φύκια. Εάν τα μεγάλα ψάρια είναι παράνο, η προστασία των, των φυκιών δεν αλλάζει. Εάν όμως φύγουμε από αυτά τα ψάρια που είναι μέσα και πάμε στα μεγάλα ψάρια που είναι πολύ πιο αρπακτικά, βλέπετε την επίπτωση. Βλέπετε λοιπόν και παραλαμβάνω υπάρχει με την, η συνέργεια που υπάρχει μεταξύ των μεν και των δε. Συμπεράντος λοιπόν όλα αυτά λέγω τα βασικά μου ευρήματα είναι τα εξής η υπερβολική υπεραλίευση συμβάλλει στην αύξηση των φυκιών η offshore λοιπόν η, ανοιχτή, η, θύρευση, η υπεραλίευση η οποία γίνεται στην ανοιχτή θάλασσα επίσης συμβάλλει σε αυτό το θέμα και κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει και το έχουμε πειραματιστεί βλέπετε αυτό το οποίο υπάρχει και το οποίο είναι το πιο σημαντικό σε αυτή τη θάλασσα ότι πρέπει και επικρατεί ο γάδος. Μόνο έτσι υπάρχει μια ισορροπία. Ιδιαίτερα στις παράκτης περιοχής. Αυτά είχα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστούμε, Δόκτωρ Έριξον, και για να ολοκληρώσουμε, Δόκτωρ Μπραντ Ντεγιάνγκ από το Πανεπιστήμιο Μεμόριαλ του Καναδά, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις ε, απαντήσεις ε, σε όλη φορά τη διαχείριση αυτών των ζητημάτων και προβλημάτων. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να ξεκινήσω ε, βλέποντας τον ορισμό σχετικά με τις αλλαγές καθεστώτος στα θαλάσσια οικοστήματα που είναι απότομες αλλαγές ε, στα οικοστήματα. Ο λόγος, το ερώτημα είναι γιατί μας ενδιαφέρει. Πρόκειται για ένα επιστημονικό ζήτημα ή ένα ζήτημα που αφορά στην διαχείριση των θαλασσών. Αφενός θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το απότομη αλλαγή και αυτό είναι δύσκολο να, ε, σε αυτό είναι δύσκολο να απαντήσουμε άμεσα και ε, υπάρχει παράλληλα και αιμονή ε, στις αλλαγές αυτές ε, του καθεστώτος. Και κάτι το οποίο θα σας μιλήσω είναι ότι περιμένουμε συνεχείς αλλαγές. Λοιπόν, αυτή η συχνότητα των αλλαγών που μας Αυτό που υπόθηκε νωρίτερα είναι ότι χρειάζεται ανθεκτικότητα. Η ανθεκτικότητα είναι το χαρακτηριστικό κάθε συστήματος προκειμένου να αντιστέκεται σε αλλαγές. Αν μειωθεί λοιπόν η ανθεκτικότητα του θαλασσίου οικοσυστήματος, τότε μειώνουμε και την δυνατότητα ανταπόκρισης στις αλλαγές. Εδώ στην διαφάνεια έχουμε ένα οικοσύστημα στο αριστερό τμήμα. Δεν λειτουργεί εντάξει. Αριστερά πάντως έχετε ένα σύστημα που είναι σχετικά ανθεκτικό και εάν επιβάλλουμε αλλαγή στο σύστημα με την ανθεκτικότητα που έχει δεν θα το τροποποιήσουμε αλλά αν μειωθεί η ανθεκτικότητα τότε θα ε, αλλάξει και το οικοσύστημα. Θα σας αναφέρω μερικά παραδείγματα σχετικά με την ε, και θα μιλήσουμε για τα χαρακτηριστικά και θα προσπαθήσω να εστιάσω στα θέματα της ανθεκτικότητας, των αβεβαιότητας ό,τι φορά την κατανόηση, την ανταπόκριση, την απάντηση και πώς θα μπορούσαν όλα αυτά να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο μιας διαχείρισης. Υπάρχει αρκετή αβεβαιότητα στο ζήτημα της διαχείρισης των αλλιευμάτων τώρα. Σε ό,τι αφορά τους κοραλογενείς υφάλους τώρα, να πω ότι υπάρχουν κάποιε διαφοροποιήσει, αλλά, αλλά σε ό,τι φορά του ωκεανού, τα πράγματα είναι διαφορ, ήταν διαφορετικά. Από το 1990 μέχρι το 2000 ε, υπήρξε διαφωνία αναφορικά με το κατά πόσον ήταν γεγονό ότι αυτό αλήθευε αναφορικά με τους ωκεανούς. Τώρα, για τα κορολογιονείς υφάλους, οι ε, αλλαγές στο σύστημα και στην ουσία αυτό το οποίο συνέβη ήταν μια μετατόπιση της, ε, της ε, μια αύξηση τους, μια αποδυνάμωση μάλλον των δυνατοτήτων των κορολογικών υφάλων. Και ένα από τα προβλήματα ήταν ε, αυτό των αχινών. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν τα οποία ε, οδήγησαν σε αυτή τη μετατόπιση, αυτή την ε, κατάρρευση, ήταν η διαχείριση των κοραλιογενών υφάλων και με την αφαίρεση των αλλιευμάτων βλέπουμε αυτήν την δραματική αλλαγή σε ό,τι αφορά την αύξηση των φυκιών στις, στους καλογενείς και βλέπετε λοιπόν την ε, μετάβαση από ένα υγιές σε ένα μη υγιές σύστημα. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρέασαν τους κορολογικούς υφάλους όπως το ζήτημα της ε, ακτινοβολίας, ε, το φόσφορο, ενεργή του φωσφόρου, τον, του, του συγγνώμη το ύδατος. Υπάρχει ένα άλλο παράδειγμα από τον ειρηνικό που ανέφερε ο Κρίστιαν νωρίτερα. Από το 70 μέχρι το 90 το τι έγινε, ποιες αλλαγές υπήρξαν. Έχουμε εδώ εικόνες για τα αλλιεύματα και βλέπουμε ε, ότι υπήρχε μετάβαση σε ένα σύστημα το οποίο, ε, το οποίο κυριαρχούσαν ε, οι χθείς ε, όπως το γάδος του Βορρά οι γαρίδες και τα σπόνδυλα γενικότερα αυξήθηκαν. Μπορείτε να δείτε επίσης πως ε, τα, όλα τα είδη δεν μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα ή ταυτόχρονα. Υπάρχουν ε, ε, εχθείς που ανταποκρίνονται πιο γρήγορα, ε, με μεγαλύτερη καθυστέρηση. Τώρα, η ιδέα μου αναφορικά με το θέμα της ανθεκτικότητας ε, και το τι συμβαίνει όταν ε, υπάρχει υπεραλίευση στους κορολογινούς υφάλους ε, συχνά υπάρχει μια μείωση της ανθεκτικότητας μετά από ρελεύση και έτσι γίνονται πολύ πιο ευάλωτοι σε εισβολείς Έτσι το όλο σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ε, ανάγκες και έτσι οδηγούμεθα σε μια αύξηση των ε, φυκιών και καταστρέφεται το οικοσύστημα των κοραλιογενών υφάλων. Και όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ πιο εύκολο και απλό να καταστρεφεί κάτι παρά να αναδομηθεί και να επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση. Ένα από τα χαρακτηριστικά της περιπλοκότητας αυτών των οικοσυστημάτων είναι πως ε, δεν ε, γνωρίζουμε πού ακριβώς πηγαίνουν, πώς ε, πηγαίνουν και η προσπάθεια να τα, να τα επηρεάσουμε είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφύγουμε. Αλλά είναι γεγονός ότι οποιαδήποτε προσπάθεια που θα έχει ως αποτέλεσμα την επαναφόραση μια προηγούμενη κατάσταση, όπως έχει συντηθεί το ζήτημα στον ε, Ατλαντικό για το ζήτημα της, ε, του γάδου. και να επανέλθει στην ε, προτεραιά κατάσταση. Λοιπόν, αν κοιτάξουμε εδώ τις συνθήκες της αρχής του 1990, και τους ε, διάφορους δείκτες που έχουμε. Εδώ μιλάμε για την περίοδο όπου ήταν ευνοϊκή η περίοδος για, την, ε, για τους ηχθείς ε, και όχι για τα ασπόνδυλα. Α δούμε λοιπόν κάποιες χρόνος σειρές, τα θηρευτές βλέπουμε ότι μειώθηκαν και με την μείωση αυτή οδήγησε σε μείωση, και εξαφάνιση των ασπονδύλων. Οι γαρίδες και τα ασπονδύλα λοιπόν επηρεάστηκαν και τα μικρά μεσαία είδη μειώθηκαν διότι οι θηρευτές αυτών των ειδών αυξήθηκαν. Έχουμε μερικά παραδείγματα τα οποία όμως είναι σαφή, υπάρχουν όμως και ενδείξεις ότι η αύξηση της θερμοκρασίας έπαιξε σημαντικό ρόλο. Τώρα αν επανέλθουμε στο σύντημα τώρα της περιπλοκότητας ε, του συστήματος, εδώ μιλάμε για μια περίοδο 30-40 ετών από το δεκαετία 60 στο 90. Βλέπουμε ότι άλλαξε η σύνθεση και έγιναν αλλαγές παράλληλα με τις αλλαγές θερμοκρασίας και έγινε και μια ανακατανομή θα μπορούσαμε να πούμε και μπορούμε να αναρωτηθούμε αν όλοι οι μικροοργανισμοί έχουν ε, το ίδιο μέγεθος. Ο λόγος για τον οποίο αυτό θα πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι ότι κοιτάζοντας την περίοδο από το 60 μέχρι το 90, η αριστερή πλευρά βλέπουμε τα, τα ψυχρά ύδατα και τα θερμά ύδατα και τους οργανισμούς που ζούσαν σε αυτά. Βλέπουμε λοιπόν ότι ε, υπάρχει αυτή η διαφορά ανάμεσα στο 60 και το 90 και έτσι οι στήλες που βλέπουμε αφορούν ε, ε, το φθινόπωρο και την άνοιξη. η αλία η οποία επηρεάζει τόσο τους μικροοργανισμούς όσο και το σύστημα στο σύνολό του, ε, αλλά έχουμε και την ε, παρεμβολή του κλίματος και των κλιματικών συνθήκων και πρωτίστως της θερμοκρασίας. Εδώ βλέπουμε κατά πόσον, ε, πόσο μάλλον επηρεάζουν οι κλιματικές συνθήκες αλλά και η αλίευση, η υπεραλίευση. Στον Βόρειο Ειρηνικό αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει μια ε, φυσική ροή των πραγμάτων, δεν μπορούμε να παρέμβουμε, είμαστε αναγκασμένοι να προσαρμοστούμε τώρα να συνοψίσω κάποια σημεία. Τα... Η μετατόπιση είναι κάτι το κοινό, κάτι το ευρύ και αφορά και το σύνολο του οικοσυστήματος. Το εντοπισμό είναι όντω δύσκολο, ε, χρειάζεται και οι κατάλληλε γνώσει, οι οποίες όμως συχνά απουσιάζουν για τα πιο περίπλοκα οικοσυστήματα είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πολλά. Τώρα η ανθεκτικότητα είναι ένα ζήτημα κλειδί και οι ανθρωπογενείς δραστηριότητε, οι ανθρώπινες δραστηριότητε ε, επηρέασαν στο να μειώσουν την ανθεκτικότητα και ενδεχόμενα να αυξήσουν τη μετατόπιση. Οι μετατοπίσεις ε, αυτές όμως ε, είναι αβέβαιο το πώς ε, θα εξελιχθούν το εδώ. Στο αριστερό τμήμα βλέπετε το ζήτημα της βιωσιμότητας και δεξιά τα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα τα κοινωνικά και οικονομικά συστήματα φαίνεται ότι βαρύνουν περισσότερο το θέμα της διαχείρισης των συστημάτων είναι κάτι πιο περίπλοκο. Είδαμε λοιπόν πως η αλληλεία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανθεκτικότητα του οικοσυστήματος μετά από ένα καθεστώς μετατόπισης ε, υπάρχει μια επιστροφή, η επιστροφή στην ε, προτεραία κατάσταση μπορεί να χρειαστεί πολύ χρόνο. Η διαχείριση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ε, όλες αυτές τις συνθήκες. Δεν υπάρχει κάποιο εργαλείο συγκεκριμένης για κάποια αντιμετώπιση της, ε, ε, του μετατόπιση των συστημάτων. Οι μετατοπίσεις όμως ε, των οικοσυστημάτων στους ωκεανούς είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ενταχθεί στην διαχείριση των υδάτων και των αλλιευμάτων. Και τέλος ε, να πω ότι χρειάζεται ένα παγκόσμιος ε, προγραμματισμός Η ανθεκτικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό και το οποίο θα πρέπει να προσδιορίσουμε και να μετρήσουμε με καλύτερα το μετώπιση καθεστώτων απαιτούν διεθνή συνεργασία διότι συμβαίνουν, αυτά που συμβαίνουν στον Βόρειο Ατλαντικό μπορεί να επηρεάσουν και τον, ε, τις θάλασσες του Νότου. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα λοιπόν δεν είναι σίγουρο ότι θα ε, το βρούμε μπροστά μας ε, και αργότερα. Ευχαριστώ πολύ δόκτωρα Γιάνγκ και τώρα έχουμε 34 λεπτά στη διάθεσή μας ε, για συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους ομιλητές. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Επί μια μισή ώρα σας ακούσαμε και τα έγγραφα τα οποία έχουμε αναχείρας θα μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. Λυπάμαι που δεν είμαστε πολύ άριθμοι σήμερα, αλλά φυσικά το μήνυμά σας είναι τεράστια σημασία και θα χρειαστεί να το λάβουμε περαιτέρω υπόψη μας στη μεταρρύθμιση της κίνησης αλληλευτικής πολιτικής όχι μόνο για τις οικονομικές επιπτώσεις των ε, μετατοπιστών καθεστώτων, αλλά και την υποβάθμιση των ε, θαλασσίων συστημάτων. Εγώ είμαι Σουηδέζα και γνωρίζω πως τη μεγάλη τραγωδία είναι για τους Σουηδούς πολίτες να βλέπουμε να πολλαπλασιάζονται τα φύκια στην Βαλτική. Κύριε Κασίνη, μας ε, δώσατε πληροφορίες σχετικά με την γραμμική σχέση ε, της υπερλίευσης του γάδου και την εμφάνιση αυτών των ε, φυκιών. Άρα εμείς ως κοινωνία θα γνωρίσουμε τις ε, επιπτώσεις αυτής της ε, αλίας ε, και όχι μόνο οι αλίες θα την αισθανθούμε και ακόμα και στον αγροτικό τομέα διότι το ζήτημα του ευτροφισμού κοστίζει τεράστια ποσά στον αγροτικό τομέα και για όλες τις χώρες πέριξ της Βαλτικής οι οποίες δαπανούν εκατομμύρια από εκατομμυρίων ευρώ για να μειώσουν τις ε, εκπομπές ε, των ε, αυτών των θρεπτικών ουσιών για να περιορίσουν τον ετροφισμό. Τι είναι η μέτρα που λοιπόν, πιστεύετε ότι η επιστροφή των θηρευτών αυτών των εισβολέων στην Βαλτική θάλασσα θα μπορούσε να επηρεάσει τον ευτροφισμό. Λαμβάνει υπόψη και τις ε, εκπομπές από πλευράς γεωργία, αλλά και τα γεωργικά απόβλητα. Έχω πολλές ερωτήσεις. Η μία Κοιτάξτε, όλοι μιλήσατε για ε, μια καλή κατάσταση του θαλάσσιου οικοσυστήματος που θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει περαιτέρω πιέσεις όπως ε, το κλίμα, τα αλόχθωνα είδη κλπ. Εμείς τώρα συζητάμε τη μεταρρύθμιση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής ε, για να έχουμε κάποιους στόχους αναφορικά με την διαχείριση των εμπορικών ε, ε, ηχθείων σε επίπεδο MSY μέγιστη βιώσιμη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τις απόψεις σας. Πιστεύετε λοιπόν ότι είναι επαρκής η ανθεκτικότητα προκειμένου να διατηρηθούν τα αλλιεύματα σε αυτή τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. και όλα αυτά λαμβάνουν υπόψη τις αλλαγές του κλίματος, ε, τα αλόχθωνα είδη, ε, τις πετρελοκυλίδες ε, και ούτω καθεξής. Τώρα, συστήματα έγκαιρης προειδοποίηση, το θίξατε. Μιλήσαμε επίσης για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και τη της. αλλά στην ουσία δεν είναι εφαρμοστικό. Λοιπόν, ε, το σύστημα έγκαιρη προειδοποίηση θα μπορούσε να λειτουργήσει ώστε να επηρεάσει την διαχείριση των αλλιευμάτων. Και μια τεχνική φύση ερώτηση τώρα για τη βιομάζα. Ο ευτροφισμός αυξάνει την βιομάζα Ποια είναι η σχέση μεταξύ του όγκου των αλλιών και του όγκου του φυτοπλακτών γενικά στην Βαλτική και την Μαύρη Θάλασσα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που είπε ο Δόκτωρ Κασίνη αφορά στο, λιγό, στο μικρότερο βάρος ε, της ε, Σαρδελόρεγκας ε, και της Ρέγκας. Αλλά αυτό οδήγησε σε λεπτά, πιο λεπτά ψάρια. αλλά επηρέασε και τα θαλασσοπούλια. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στην έλλειψη βιταμίνης Β στα θαλασσοπούλια με την μείωση κάποιων βιταμινών σε άλλα είδη, π.χ. σολομό, σε άλλα θα μπορούσε λοιπόν να σου πει κάτι ο κύριος Κασίνη σχετικά. Υπάρχουν παραδείγματα σχετικά με την επιστροφή σε προτεραία κατάσταση είτε φυσικό τρόπο είτε με ανθρωπογενή παρέμβαση. Δεν ξέρω ξέχασα κάτι. Τώρα για τα μέδουσες. Τι τρώνε. Τρώνε αυγά ψαριών. Ή εδώ έχουμε κάποιο φαύλο κύκλο. το κόστος ενδιαφέρον. Ο κύριος Έριξον μίλησε για 865 εκατομμύρια ευρώ ετησίως το κόστος ε, των θικιών και 177 εκατομμύρια ε, ετησίως για την αλία. Με αυτό είναι το σύνολο του Ταμείου Αλίας. Μπορείτε να μας πείτε πώς αφορούν το τομέα της και πώς άλλους κλάδους που επηρεάζουν το, επηρεάζονται από τα φύκια. και τη διασύνδεση ανάμεσα στις κλιματικές αλλαγές και την υπεραλίευση που δεχόμενο οδηγεί σε αυτές τις αλλαγές καθεστώτος στα θαλάσσια οικοσυστήματα δείτε λοιπόν ότι αυτές οι αλλαγές, αυτές οι μετατοπίσεις θα συνέβαιναν εάν δεν είχαμε διαχειριστεί τα αποθέματα των αλλιευμάτων με τον τρόπο που το πράξαμε στη Βαλτική παραδείγματος είχαμε βάλει ως κνησιμότητα το 1,6 αντί 0,3 αυτό θα είχε μειώσει την ε, λήψη αν δεν είχαμε ε, ασκήσει λοιπόν μεγάλη ε, ε, μεγάλη πίεση στην αλλιεύματα της περιοχής. Μήπως θα είμαστε τώρα σε καλύτερη κατάσταση. Αυτά. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ε, θα κάνω εγώ μερικές ερωτήσεις γενικού χαρακτήρα και αναφέρομαι στο εξή. Γνωρίζετε πολύ καλά πως η μεταρρύθμιση της ε, κοινή ελευθερικής πολιτικής που υπάρχει επιτάπητος, η μελλοντική έρευνα έχει μια εστίαση οικοσυστημική. Τώρα η έρευνα δεν ε, έχει βασιστεί σε κάτι τέτοιο τώρα και ρωτώ επειδή διάφοροι είπατε ότι λείπουν στοιχεία στο οικοσυστημική προσέγγιση τι, τι έχετε να πείτε για το μέλλον γνωρίζοντας ε, το πώς ε, έχει η έρευνα τώρα στην Ευρώπη. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρχει μια δραστηριότητα πολυεπίπεδη. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν ποιες είναι οι δυσκολίες που βλέπετε να υπάρχουν τώρα. Και επίσης ε, εσείς ήρθατε για να μας μιλήσετε για το σύστημα, οικοσύστημα, ε, αλλά στο πλαίσιο πάντα της αλίας. Αλλά βάσει όλα τα input που έχουμε σε ένα οικοσύστημα, η αλληλεία είναι αυτό το οποίο ε, μελετάται καλύτερα πέραν των ελλείψεων που υπάρχουν και των προβλημάτων που υπάρχουν. Είπατε ότι η αλληλεία επηρεάζει το όλο σύστημα όπως ε, είναι γεγονός, αλλά η αλληλεία φυσικά επηρεάζεται από όλα τα input ε, που εισέρχονται στο οικοσύστημα. Όταν μιλάμε για οικοσύστημα, ε, γενικά ε, επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην Αλγία και λιγότερο στην ε, Γεωργία, τις μεταφορές, το κλίμα κλπ. Διότι ξέρουμε λιγότερο τις επιπτώσεις ε, από τα στοιχεία αυτά στο οικοσύστημα. Για να μπορούμε να λάβουμε λοιπόν κατάλληλα μέτρα διαχειριστικά θα πρέπει να γνωρίζουμε όλες τις αλληλεπιδράσεις και τις διαδράσεις που υπάρχουν τα, πιο ψυχρά ύδατα, έχουμε κάποιες επιρροές στην, στο γάδο κλπ. Μεθρυπήσουμε λοιπόν όλα τα input που λειτουργούν σε ένα σύστημα, τουλάχιστον βασικά από αυτά τα input, την χάνουν της αυτής γνώσης, όπως με αυτά τα οποία γνωρίζουμε στον τομέα της αλίας. Αν και στον τομέα της αλίας έχουμε λήψεις, υπάρχουν άλλοι κλάδοι για τους οποίους γνωρίζουμε ακόμα λιγότερο. Και κάποια μέτρα τα οποία λαμβάνονται, ίσως να μην έπρεπε να λαμβάνονται αν Είχαμε μια θεώρηση σφαιρικότερη του οικοσυστήματος Αυτά σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις μου προς εσάς. Ας περάσουμε λοιπόν στις απαντήσεις και να δώσω το λόγο τώρα αντιστρόφως στους προσκεκλημένοι μας πρώτα ο Δόκτωρ Γιάνγκ και μετά θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Και παρακαλώ το πολύ 5 λεπτά έκαστος, διότι σε 11 η ώρα πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό το workshop. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you, and uh, thank you for the opportunity to respond. Let me go through the question. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να απαντήσω και να εστιαστώ πολύ περισσότερο στα οποία αυτά, σας το οποία είχα πει όσον αφορά τις προκλήσεις ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι είναι αυτή η πρόκληση που υπάρχει για μία προσέγγιση του οικοσυστήματος. Μόνο έτσι. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να το πλησιάσουμε. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ισορρόπηση, Υπάρχει πληροφόρηση, αλλά υπάρχουν πολλές επι, επιρροές εάν υπάρχει το ζωοπλάνκτον, υπάρχει το φυτοπλάνκτον, πώς μπορεί να υπάρξει πραγματικά αυτή η ισορροπία, ποια στοιχεία από όλα αυτά που αναφέραμε θα λάβετε υπόψη για να υπάρξει μια εξισορρόπηση και να ακολουθήσετε ένα σχέδιο το οποίο έχει σχεδιαστεί, διότι αυτό το σύστημα του οικολογικού εξισορρόπησης εάν ε, δεν ξέρουμε γιατί το κάνουμε και το κάνουμε μόνο για σοσιοοικονομικούς λόγους, σκόλου ε, λόγους μόνο δεν αρκεί, αλλά σκοπός είναι για μας τους όπως θέλουμε να υπάρχει μια στρατηγική η οποία θα είναι ολική, σφαιρική που θα καλύπτει όλα και θα καλύψουμε, θα φτάσουμε στους τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Δεν υπάρχει βασικός λόγος γιατί δεν θα πρέπει εμείς αυτή τη στιγμή να εφαρμόσουμε αυτή την προσέγγιση που σας είχα πει. Δεν, ε, έχουμε πάντα πλήρη πληροφόρηση. Ο καιρός είναι τεράστιος, δεν μπορούμε να έχουμε όλα τα στοιχεία, αλλά και αν ακόμη ξοδέψουμε κάποια στοιχεία και εξοδέψουμε ορισμένα χρήματα, νομίζω πραγματικά δεν έχουμε καλύψει όλα τα θέματα, αλλά το θέμα της διαχείριση όσον αφορά την περιπλοκότητα όλου του οικοσυστήματα, για να πάρουμε την αλία και πάρουμε όλους τους άλλους παράγοντες εκτός, μεταφορές κλπ. γιατί σε πολλές περιοχές, ξέρετε πολύ καλά η Λυΐα είναι άλλο τομέα και άλλο τομέα είναι η μεταφορά από αλλού και από άλλους παράγοντες εξαρτώνται. Αλλά αναγνωρίζω πως όλα αυτά είναι μια πρόκληση. Όσον αφορά το σύστημα έγκαιρης προειδοποίηση είναι αυτή τη στιγμή το θέμα της ανάπτυξης να υπάρξει μια συνειδητοποίηση αυτού του καθεστώτος, αλλαγής καθεστώς που έχει γίνει και όταν υπάρχουν αυτά τα πράκτορια αυτές οι εταιρείε για τη διαχείριση της αλληλείας θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά για την υγεία και οι άλλοι προσφέρουν, όλοι οι άλλοι παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να μπουν μέσα σε αυτό το προσέγγιση του οικοσυστήματος θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να υπάρχει μια αιτήσια ή διαιτήσια ε, εκτίμηση των τεκτενομένων και όσο περισσότερο γνώση έχουμε από το θέμα του αυτού τόσο καλύτερα θα είναι και νομίζω θα είναι αυτό πολύ καλύτερο. Τώρα όσον αφορά για να υπάρξει βιώσιμη απόδοση το μάξιμο όσο ανώτερο γίνεται. Είναι καλό αυτό το πράγμα, να ένα πράγμα κανείς θα πρέπει να περιμένει. Αυτό δεν σημαίνει ότι εξασφαλίζεται κάτι. Διότι βεβαίω μειώνει τη δυνατότητα κατάρρευση του συστήματο, αλλά δεν εξασφαλίζει τίποτα. Διότι πάντοτε, πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνο μια δραματική αλλαγή του κλίματο μια θέρμανσης και βεβαίως κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξουν όλα αυτά. Αλλά εγώ δεν προβλέπω ότι κάτι τέτοιο δραματικό θα συμβεί, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτά επηρεάζουν το όλο σύστημα. Ανεξαρτήτως λοιπόν ποια στοιχεία έχουμε αναχίας, βλέπετε τι άλλαγες μπορεί να γίνει Μπορούμε λοιπόν να έχουμε το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε και να αποτελεσματικό είναι να μειώσουμε την αλίευση, διότι η υπεραλίευση δημιουργεί πρόβλημα. Και μακροπρόθεσμα θέλουμε να αυξήσουμε το καθαρό εισόδημα, το καλό το οποίο μπορούμε να πάρουμε από τον ωκεανό θα νομίζω πως σταματάω εν ευθέτω το χρόνο και δεν το δώσω στον επόμενο. Ο, ο Έριξον, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις που έτσι θα ξεκινήσω με το θέμα του κόστους. Δεν είμαι οικονομολόγος βεβαίω, αλλά τα στοιχεία της από την έκθεση της Εκκομισιόν που έχει γίνει όσον αφορά τα φύγια και τις επιπτώσεις στο οικονομικό επίπεδο. Δεν καλύπτει όλη την Ευρώπη βεβαίως και δεν καλύπτει Μεσόγειο ασφαλώς. Αλλά τα περισσότερα από αυτά αυτή τη στιγμή έρχονται από τον τουρισμό. Μετά είναι το εμπορική αλίευση υπάρχει ε, περιεχόμενο το πρόβλημα της παρακολούθησης. Η Σουηδία, για παράδειγμα, γνωρίζει πολύ καλά αυτό το θέμα. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν πολλά. Φύγε εκεί. Και αυτό είναι ένα κόσμο που Επίσης έχει ένα κόστος στην ανθρώπινη υγεία, όταν οι άνθρωποι αρρωσταίνουν γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να έχεις κακά στρίδια. Αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να είμαστε σε θέση να υπάρξει ένα σύστημα, μια καλή διαχείριση του οικοσυστήματος. Καθώς, μπράβο. Η προτασιμότητα είναι ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό. Είναι μια το οποίο έχουν κάνει πολλοί επιστήμονες από διάφορα πανεπιστήμια, από οργανισμούς, διότι είναι αδύνατο να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Το προσπαθήσαν πολλές φορές. Και αυτό ισχύει για πολλές χώρες βεβαίως τα συμφέροντα, τα οποία είτε είναι ιδιωτικά, είτε είναι διάφορων ε, οργανισμών κλπ. Το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το σημείο είναι ότι όλα είναι προσβάσιμα η αύξηση των θηρευτών ψαριών είναι πολύ καλύτερη και ποια είναι η επίπτωσή του σαν αφορά τα φύκια. Είναι θέμα δύσκολο αυτό. Οι θηρευτές όταν φύγουν οι θηρευτές δεν αυτομάτως δεν ευεργούνται τα φύκια, αλλά υπάρχει μια πίεση η οποία δημιουργείται. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν είναι μια δεν είναι ελληνική λύση, αλλά είναι μια συμπληρωματική λύση η οποία μπορεί να βρεθεί. Αυτό το οποίο όταν υπάρχει περισσότερο ευστροφισμός έχετε πάρα πολύ καλά στοιχεία τα οποία έρχονται από την Βαλτική, από την Ολλανδία κλπ. Αλλά δεν είχαμε τις απαντήσεις αυτές οι οποίες θα προσμέναμε να έχουμε. Μπορεί να με διορθώσετε αν εσείς έχετε διαφορετική άποψη, άποψη κύριε συνάδελφοι. Το τελευταίο θέμα έχει σχέση το, τη βέλτιστη βιώσιμη απόδοση το, ή τη μέγιστη. Έτσι λοιπόν πιστεύω πραγματικά ότι έχουμε την μέσα εκείνα μέτρηση για να δούμε πού μπορεί να είναι αυτή η μέγιστη πρέπει να σκεφτούμε ποιο είναι το μάξιμο σε ένα, μέσα σε ένα οικοσύστημα. Είναι ένα θέμα περίπλοκο και πολύπλοκο και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλα συνδέονται μεταξύ και δεν είναι μόνο ποιο, πόσα ψάρια παίρνουμε πέσα από αυτόν τον πληθυσμό, αλλά υπάρχουν και άλλοι οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να δοθούν και βεβαίως και αυτοί πλήττονται. Πλήττονται ιδιαίτερα στη Μαύρη Θάλασσα όταν έχουμε αυτά τα προγράμματα. Στο τέλος πραγματική θα πρέπει να δούμε πώς θα υπάρξει μια ισορρόπηση μεταξύ αυτών των πραγμάτων και όχι μόνο για τους παραγωγούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο καθηγητής Δασκάλοφ έχει το λόγο, παρακαλώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας με μια θετική άποψη. Ναι, πραγματικά αυτό που είπατε πραγματικά συμβαίνει και αυτό συμβαίνει ενίοτε χωρίς να γίνεται κάποια διαχείριση όλο στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτή η αλλαγή που γίνεται μπορεί να δώσει τη δυνατότητα μια ανάρρωση. Υπάρχει μια βέβαια υπάρχει μια καταστροφή που έγινε εκεί, μια πτώση η οποία είναι εκατομμύ... δεκάδες εκατομμύρια. Τρία χρόνια έχουμε καλύτερες οικολογικό περιβάλλον και για τα αποθέματα και την αύξηση των ψαρών, ιδιαίτερα στο τη χαμηλή αλίευση. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο στον ευξηνοπόντο, αλλά και η αλληλεία μειώνεται λόγω της έλλειψης αποθεμάτων δυστυχώς. Σε τέτοιες περιπτώσεις βεβαίω. στο σύστημα αυτό καθ' αυτό είναι πολύ τροτό η επιδείνωση των καιρικών συνθήκων βεβαίως έχει την επίπτωσή της καθώς επίσης η εισβολή ορισμένων ειδών ένα, ένα γαστρόποδο κεφαλόποδο το οποίο έχει, έχει έρθει στη Μαύρη Θάλασσα όλα αυτά τα ξένα ψάρια και είδη μπορούν να εξορροπήσουν μέχρι σε ένα σημείο, να μέχρι στιγμή, μέχρι κάποια στιγμή, αλλά μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα και βεβαίω οι δραματικέ αλλαγέ όπω η αύξηση θερμοκρασία είναι πάρα πολύ επί παράγοντες και βλαπτικοί παράγοντες. Υπάρχουν και άλλα συν και σε άλλα πράγματα βλέπουμε ότι το σύστημα μόνο του αυτορυθμίζεται. Υπάρχει όμως μία τάση να πάμε στην, σε μία καλύτερη κατάσταση ή να φτάσουμε στην παλαιότερη κατάσταση, αλλά πιστεύω πως Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή τη διαχείριση να του βοηθήσουμε και θα ήταν οι πάντε θα ήταν ευτυχέστεροι αν υπήρχαν οι καλύτερε συνθήκες και θα μπορούσαμε τελικά να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την πίεση. Διότι ξέρετε υπάρχει όλη αυτή η πίεση η οποία έρχεται από το περιβάλλον, όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε προαναφέρει και τα οποία είναι οφείλεται σε ανθρώπινους παράγοντες, σε φυσικούς παράγοντες και οι οποίοι επιδρούν. Νομίζω λοιπόν σκοπός είναι αυτή τη στιγμή το σύστημα να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή θέση και κατά κάποιο τρόπο είναι σωστό να υπάρχει αυτό διότι υπάρχει, όπως ξέρετε, πάρα πολύ καλό και ένα θέμα εφαρμογής, εφαρμοστικότητας όλων αυτών των πραγμάτων. Βεβαίως, εάν θέλουμε πραγματικά να αποτιμήσουμε ποια θα είναι η επίπτωση στο όλο οικοσύστημα, θα πρέπει να ακολουθήσουμε μοντέλα τα οποία θα είναι πολύ πιο περι, πρότυπα, πολύ πιο ε, περίπλοκα, όπως το και Καθώς όλα αυτά επιδρούν. Το MSY είναι πολύ διαφορετικό για διάθε είδος και για κάθε απόθεμα. Όσον αφορά λοιπόν τη διαχείριση, η παρούσα κατάσταση είναι πολύ καλή εάν, την, εάν επιτευχθεί. Βεβαίω μπορεί να υπάρξει βελτίωση σε αυτήν την κατάσταση για το πλανκτόν και για το οικοσύστημα αυξάνεται πάρα πολύ το πλακτόν γιατί εγκαταλείφθηκε. Αναφέρεται επίσης Κατά την άποψη μου δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό το τελευταίο σημείο που σας ανέφερα, αλλά υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι ε, συμφωνούν ότι είναι σημαντικό. Υπάρχει όμως μία επίπτωση σε όλη τροφική αλυσίδα μέσα από αυτά τα πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο καθηγητής Καζίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα προσπάθησω να απαντήσω μερικές αυτέ τι ερωτήσει και πιστεύω πως το θέμα κατά πόσο η διαχείριση της αλλίευση είναι πολύ πιο αποτελεσματική, είναι πιο αποτελεσματική παρά και η μείωση των, διατροφι θρεπτικών στοιχείων. Αλλά πιστεύω και συμφωνώ πως η διαχείριση της, του αλλιεύματος μπορεί να συμβάλλει πολύ βεβαίω στη μείωση της αύξησης των φυτιών. Αυτό το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε και να διάνουμε είναι τα απλούστερα προβλήματα τα οποία δεν προσπαθούμε να ιάσουμε τα βασικά πράγματα. Αυτό είναι μία πηγή. Η άλλη είναι οι εκπομπές. Αυτό είναι ο λόγος για πιστεύω πως θα πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές, στην ένταση των εκπομπών και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συγκρατήσουμε αυτές τις εκπομπές εν πάση περιπτώσει. Ωστόσο, η μείωση του αλλιεύματος νομίζω πως πραγματικά θα μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ καλό συμπληρωματικό μέτρο σε αυτό, γιατί θα, θα υπάρξει αυτή τη στιγμή μείωση πολλών συμπτωμάτων τα οποία ανακύπτουν και φαίνεται αυτό το τελευταίο διάστημα. Όσον αφορά το θέμα του MSY, το MSY όπως ξέρετε είναι μόνο για τα εμπορικά είδη εκείνα των ψαριών δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι αυτά τι επίπτωση έχουν στη χαμηλή διατροφική αλυσίδα. στον είναι ο λόγος για τον Αυτή η προσέγγιση έχει σαν σκοπό να έχει μία ελίευση σε ένα ορισμένο επίπεδο με παράλληλα με, με, υψηλή, με υψηλό βαθμό αλίευσης. Συνεπώς, αυτή η προσέγγιση δεν είναι πολύ συνεκτική με μία ε, προσέγγιση η οποία θα ήταν πλήρως, πλήρως οικοσυστημική. Έτσι λοιπόν θα προσπαθείς γίνεται να γίνει αλλαγή αυτής της προσέγγισης μόνο για ένα είδος και γίνεται μια προσέγγιση η οποία θα είναι για πολλά είδη και για την προστασία του βεβαίω. Αλλά υπάρχει, θα πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη και νομίζω πως πραγματικά μπορεί να έχει κάποια επίπτωση επί του νομοθέτη. Θα πρέπει να απαντήσω ακόμη αυτό το θέμα της μείωσης του Σαρδελό Ρέγκας. Αυτό γίνεται και λόγω της κλιματικής αλλαγής και φαίνεται πως ε, το, η μείωση του βάρους τους επίσης έχει επίπτωση και στην αλληλεία κατευθείαν, διότι σημαίνει ότι τα λιεύματα είναι πολύ μικρά ψάρια και θα πρέπει για να καλύψουν την ποσόστοσή του να ψαρεύουν και να λιεύουν όλο και περισσότερα ψάρια. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω ωστόσο είναι ότι το γεγονός, η επίπτωση που έχει στα ψα, ε, θαλασσοπούλια και στο Σολομό φαίνεται σχετίζεται με αυτή την, τον πληθυσμό της Σαδελόρεγγας. Και υπάρχουν στατιστικές οι οποίες δείχνουν τελευταία για τον Σολομό, για, παρεμβάνω, για τον Σολομό, ο οποίος εξαρτάται από αυτόν και ε, το σύνδρομο το οποίο δημιουργείται οφείλεται σε αυτή την αλυσίδα που παρέφερα προηγουμένω. Όσον αφορά τα θαλασσοπούλια φαίνεται πως όταν αυξάνονται οι σαρδελόγγες αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό για τα θαλασσοπούλια. Εάν επανέλθουμε στο παλαιό καθεστώς λοιπόν μπορεί να είναι επιβλαβές και επιζήμιο μάλλον για ορισμένα είδη. Λοιπόν, οι πολιτικέ αποφάσει οι οποίε θα πρέπει να, να θα ληφθούν θα πρέπει να τα λάβουν όλα αυτά υπόψη. Τι ακριβώ πρέπει να αποφασίσουμε και ποιου θα ευνοήσουμε. Και ένα ακόμη πολύ σύντομο πράγμα, όταν μιλάμε για αυτά τα καθεστώτα αλλαγή, θα πρέπει να πω ότι υπάρχουν πολλέ χώρες με πολλά διαφορετικά συμφέροντα. Υπάρχουν χώρες οι οποίοι θέλουν ψηλές ποσοστώσεις για το ένα ψάρι ή για το άλλο ψάρι. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε για να χαράξουμε μια πολιτική. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο εγώ σαν τον τελευταίο ομιλητή, αλλά είπατε προηγουμένω όταν υπάρχουν αλλαγέ θα μπορεί να γίνει μια πρόληψη όσον αφορά τη διαχείριση. Υπάρχουν, ξέρετε, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο είναι πάρα πολύ υγιέ. Μπορείτε να δείτε λοιπόν ποιε είναι οι επιπτώσει. Η ενδο οργανικές επιπτώσεις είναι λιγότερες και αν πραγματικά έχετε ένα σύστημα το οποίο προλαμβάνει αυτές τις καταστάσεις δεν θα υπάρξουν αυτές τις καταστροφικές εικόνες οι οποίες σας ζώθησαν για όσον αφορά την αλλαγή αυτό του συστήματος θα πρέπει να είναι προληπτικό και με τελική αναλύση να είναι τα προγράμματα τόσο δραστικά για να μπορεί πραγματικά να προλάβουμε αυτή την πτώση αυτού του συστήματος. Επίσης το θέμα της επιστροφής. Η Βαλτική είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, διότι υπάρχουν επιστροφές σε αυτές τις περιοχές και μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει μια διασύνδεση, ένα συνδυασμός υψηλού υψηλού βαθμού διατήρησης και βεβαίως αυτό έχει μια πάρα πολύ καλή επίπτωση και στην αλληλεία και το όλο οικοσύστημα και βεβαίως μπορεί αυτό να οδηγήσει σε μια ανάρρωση αυτής όλης της κατάστασης. Και πιστεύω πως αυτό είναι το ίδιο, ο ίδιος μηχανισμός ο οποίος θα ισχύει και αυτό. Αυτή θα επανέλθω τώρα στις πρόκληση όσον αφορά αυτό του οικοσυστήματος και της προσέγγισης του οικοσυστήματος. Γιατί όλο αυτό το σύστημα έχει σχέση με την ένταξη, με την ενσωμάτωση που πρέπει να γίνει στο όλο συστομάτικο. Νομίζω πως αυτό το σύστημα είναι πολύ καλό ότι θα και μέσα δι' αυτού του συστήματος θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, να δούμε τους διάφορους τομείς, πώς πραγματικά αυτή μπορεί να λειτουργήσουν και οι διάφορες χώρες οι οποίες εμπλέκονται σε αυτή την προσπάθεια ξέρετε πρέπει να δούμε την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί και κατά πόσο πραγματικά κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε και υπάρχουν ξέρετε υπάρχει ένα Ινστιτούτο που προτείνει κάτι αλλά υπάρχουν πάρα πολλά Ινστιτούτα πολλά εμπλεκόμενοι και αυτά είναι πραγματικά εμπόδιο όσον αφορά αυτή την προσέγγιση του οικοσυστήματος και είναι και πολύ ακριβό γιατί θα πρέπει να παρακολουθούμε πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα από ό,τι κάνουμε μέχρι σήμερα, μέχρι τούδε. Και νομίζω πως αυτό είναι αρκετή απόδειξη όσον αφορά την ανιχνοσιμότητα που κάνουμε όχι μόνο για τα ψάρια για τα λέει της θαλάσσης και πιστεύω αυτό που είναι σαφές για να έχετε πραγματικά ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης θα πρέπει να έχετε πολύ σταθερά και πολύ αξιόπιστα στοιχεία τα οποία έρχονται δεδομένα βεβαίως πράγμα το οποίο κοστίζει. Αυτά είχα να πω. Σα ευχαριστώ. Νομίζω ότι μα ε, διευκρίνησατε κάποια ζητήματα που μας ε, απασχολούν. Ευχαριστώ λοιπόν όλους σας. Ε, και ευχαριστώ και την αρμόδια υπηρεσία που οργάνωσε αυτό το workshop ότι δεν ήμασταν πολύ άριθμοι οι παρεμβάσεις όμως που ακούστηκαν ήταν πολύ ενδιαφέρουσες στο σημείο αυτό λοιπόν ολοκληρώνεται το σημείο 8 της ημεστές διατάξεως και περνάμε στο υπαριθμό 9 Πρόκειται για την κοινή ελευθερική πολιτική, η κυρία Ρόντους, θα δώσω το λόγο στην κυρία Ρόντους. Ja, vielen Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σε όλη τη διάρκεια της ακρόασης. σε μια Επιτροπή όπου διεξήχθησαν ψηφοφορίες. Πάντως άκουσα το τελευταίο κομμάτι της ακροάσεως και κατάλαβα ότι όντως ήταν ενδιαφέροντα αυτά που ακούσατε. Δυστυχώς ε, δεν μπορούμε να κλωνοποιηθούμε. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν ε, μια ε, τρεις λόγους να βρούμε για τις απορρίψεις πρώτα απ' όλα. Ήδη για τα οποία δεν υπάρχουν ποσοστώσει και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο μπορούμε να προβλέψουμε κάποιες εξαιρέσεις. Ε, μετά υπάρχουν οι απορρίψεις ε, που μπορούν να περιοριστούν μέσω καλύτερη διαχείριση. Και τέλος, τα παραδείγματα και των γόνων ορισμένα ε, ήδη θα πρέπει να απορρίπτονται στην θάλασσα. Αυτό είναι ζήτημα δύσκολο. Το συζητήσαμε χθε με τον Στίβενσον και την έκθεσή του αναφορικά με την αξιοποίηση π.χ. άλευρα ε, ηχθείων και ο Αλιεύς ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει, ότι ζητάει να έχει την καλύτερη δυνατή προσφορά για τα προϊόντα του. Το, ένα σημαντικό ποσοστό των αλιευμάτων ε, ε, μετά απορρίπτονται στη θάλασσα. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Όλοι συμφωνούμε για το ότι χρειάζεται να ε, αυξηθεί η επιλεξιμότητα ε, λοιπόν, μια απαγόρευση των απορριμψέων νομίζω ότι δεν είναι το καλύτερη λύση διότι δημιουργεί δυσκολίες στους αλληλεί. Οι αλληλεί δεν γνωρίζουν ποια είναι η ποσότητα των παραδειγμάτων. Γι' αυτό λοιπόν είναι δύσκολο να γίνει κατανομή των ποσοστώσεων. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις ε, χρειάζεται να ε, υποδεχθούν αυτά, τα, αυτές τις απορρίψεις, αλλά οι δυνατότητες αυτές είναι περιορισμένες. Πολλές τα σκάφη είναι μικρά. Ε, και ιδιαίτερα στην Μεσόγειο είναι πιο οξύ το ζήτημα λόγω των μικρών αληθικών σκαφών. Τώρα, η απαγόρευση των απορρίψεων δεν είναι λύση, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε. Το status quo ούτε και αυτό αποτελεί λύση. Θέλουμε να έχουμε έναν δεσμευτικό στόχο που να συμπεριληφθεί στον κανονισμό, διότι διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βελτιώσουμε την επιλεξιμότητα των ε, εργαλείων ε, αλίευσης ε, των ελεκτικών εργαλείων. Θα πρέπει λοιπόν στον κανονισμό να θέσουμε κάποιον συγκεκριμένο και σαφή στόχο. Και κατά την άποψή μου αυτός ο στόχος θα πρέπει να είναι απαγόρευση απορρίψεων, προλέποντας κάποια εξαίρεση για τη Μεσόγειο, αλλά ε, θα πρέπει να υπάρξει μαζική μείωση αυτών των απορρίψεων. Όσοι υποστηρίζουν πως ε, θέλουν να επιτύχουν το στόχο αυτό προοδευτικά, τους λέω ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε αν αποφασίσουμε να το αναβάλουμε, να το μεταθέσουμε στις ρωμαϊκές καλένδες. Νομίζω ότι δεν θα δείξουμε την δέουσα σοβαρότητα. Φυσικά τα μέτρα θα πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν. Χρειάζεται μια οικονομική στήριξη από πλευρά ε, ταμείου. Παράλληλα, χρειάζεται και μια μεταβατική περίοδος ε, λογική και ε, ο όρος απαγόρευση καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί προβλήματα. Πρέπει να εξηγήσουμε στους αλληλείς ότι θέλουμε να τους βοηθήσουμε στην πράξη και να τους δείξουμε ότι και αυτοί θα ωφεληθούν από την λήψη παρόμοιου μέτρου. Οι αλληλείς που αλλιεύουν λιγότερο μπορούν να ε, να εκφορτώνουν στο λιμάνι ε, τις ίδιες ποσότητες. Τώρα, για τα παραλιεύματα, το ζήτημα είναι να γνωρίζουμε αν αυτό θα περάσει μέσα από τον βασικό κανονισμό ή μέσω κάποιου άλλου νομοθετήματος. Επίσης, το ζήτημα των ποσοστώσεων και ο επιμερισμός αυτών. Κάθε αλλιάς ε, θα πρέπει να λαμβάνει τις ποσότητες, τις ποσοστώσεις, συγγνώμη, που είναι απαραίτητες μια σφαλμένη κατανομή των ποσοστώσεων νομίζω δεν θα ήταν η καλή λύση. Εξού και ερώτηση προς την Κομισιόν. Ε, σε ποιο μέτρο στην πρότασή σας εγγυάστε ότι στους αλείς θα χορηγηθούν οι, ε, καλέ, οι σωστές ε, ποσοστώσεις. Λοιπόν, πώς θα λάβουν τις ποσοστώσεις αυτές οι αλίες, διερωτώ με θα ήταν προτιμότερο να ε, εισαχθεί μια εθνική ποσόστοση και όχι μια ποσόστοση για κάθε αλία. Τώρα πώς ε, θα πετύχουμε κάθε κράτος να λάβει την ε, σωστή ποσόστοση. Οι ποσοστώσεις χορηγούνται με ιστορικούς, ε, σύμφωνα με ιστορικούς λόγους ε, και τι συμβαίνει όμως αν ε, κάποια κράτος δεν θέλει να αλλάξει τις ποσοστώσεις. Μπορούμε να επιβάλλουμε αυτή την αλλαγή. Και κάτι ακόμα. Τα κράτη-μέλη θα φροντίσουν να επιλύσουν το πρόβλημα στο των ποσοστώσεων ίσως ε, θα πρέπει μέσω του άρθρου 16 να δεσμευτούν τα κράτη-μέλη ώστε να διατηρήσουν στον διαπραγμάτευση τάκ και ποσοστώσεις κάποιες ε, ποσότητες. το το θέμα της ε, επιλεξιμότητας Εδώ θα πρέπει να εφαρμόσουμε κάποιες ε, παρενέσεις, παροτρήσεις. Ε, οι αλλιείς ε, θέλουν να ζήσουν από το δουλειά της και δεν είναι πρώτο το, τους μέλημα η προστασία του περιβάλλοντος. Οι αλλιείς προτιμούν φυσικά τα ενήλικα ψάρια και όχι τον γόνο ή τα εκτίδια. και θα ήταν ε, εύλογο για τον γόνο ο οποίος αλλιεύτηκε να προβλεφθούν ποσοστώσεις υψηλότερες ε, και έτσι να ε, και παράλληλα να ενθαρρύνουμε την επιλεκτικότητα. Αυτό δεν θα οδηγήσει τους αλείς για περισσότερα παραλιεύματα, αλλά θα τους οδηγήσει στο να αποφεύγουν ε, την ε, αλίευση γόνου, γιατί φυσικά υπάρχουν ποσοστώσεις υψηλότερες για τους αλίες σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν τι έχει να μας πει η Κομισιόν και περιμένω και τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Κύριος Ρωμέβα. Πρώτα οι βουλευτές και μετά η Κομισιόν. Κύριε Ρωμέβα, έχετε το λόγο. Να ευχαριστήσω φυσικά τη συνάδελφο Ρόντους του. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά το μας είπε. Το, το πρώτο θέμα είναι το εξή. Απαγόρευση των απορρίψεων θα πρέπει να είναι ένα μέσο, αλλά εν πάση ο τελικό στόχο δεν είναι με κάποιο τρόπο να νομιμοποιήσουμε τις απορρίψεις, αλλά να αποφύγουμε την ε, δημιουργία τους. Άρα να υπάρχουν μηχανισμούς που θα αποφεύγουν το να ε, ε, υπάρχει παραλίευση. Αυτό είναι ο τελικός στόχος. Και ο κίνδυνος που βλέπω εγώ με την πρόταση της Κομισιόν είναι πως ξεχνάει τον τελικό στόχο και επικεντρώνεται ως μέτρο το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μία συγκάλυψη αλλά και θέλει να πετύχει την απαγόρευση της απόρριψης. Εδώ είναι το πρόβλημα. Κανείς ε, δεν μπορεί να φλή απέναντι σε μια τέτοια πρόταση. Ο κοινός στόχος είναι να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά ο μηχανισμός είναι αυτός ο οποίος μας ε, προκαλεί κάποιες Υπάρχουν ποικίλε προτάσεις, ε, μερικές τις ανέφερε η τις ε, τροποποιώ ή τις ε, υπογραμμίζω. Πρώτον, να καταβληθούν προσπάθεια για ε, χρησιμοποίηση αλληλευτικών εργαλείων πιο επιλεκτικού χαρακτήρα, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία και να, τα, οποία είναι πιο επιλεκτικά, κάνουμε μεγαλύτερη επιλογή των ειδών και του μεγέθους και εδώ θα πρέπει να ε, μην ασχοληθούμε μόνο με απορρίψεις που έχουν εμπορικό, εμπορικό αποτέλεσμα, αλλά και με τις άλλες απορρίψεις που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα, αλλά έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο οικοσύστημα. Επίσης η κυρία Ρόντους είπε και θέλουν να το τονίσουμε αυτό, αυτή η διάσταση των οι διαστάσεις των αντιδημάτων θα πρέπει να μας οδηγήσουν στο να ασχοληθούμε με τα αλλιεύματα γενικότερα και όχι με συγκεκριμένα είδη αλλη, αλλά και κάτι ακόμα, να υπάρχουν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις αναφορικά με τη διαχείριση αυτών των απορριμμάτων, στο μέτρο που αυτοί ε, εντάσσονται, συμπεριλαμβάνονται στην αγορά, ή να έχουν μηχανισμούς ε, ποιότητας ε, για την υλοποίηση πιο αυστηρών ελέγχων και να αποτρέψουμε την χρήση εργαλείων μη επιλεκτικών. Αυτά είναι σημεία που δεν είναι σαφή στην πρόταση της Κομισιόν. Περισσότερο από ζήτημα φόρμας τύπου είναι ζήτημα εστίασης και κινδύνου που θα πρέπει να περιορίσουμε. Μη προτάσεις πάντως που υποβάλλει η εισηγήτρια και μερικές ακόμα που θα προσθέσουμε θα μπορούσε να έχει καλό αποτελέσμα. Ευχαριστώ κύριε Στίβενσον, παρακαλώ να είστε σύντομοι διότι 12 παραθέας πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ και ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Ρόντας για όλη τη δουλειά την οποία έκανε πάνω σε αυτόν τον βασικό κανονισμό, τον κανονισμό βάσης. Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα πολλές από τις παρατηρήσεις που διατυπώσατε αλλά νομίζω ότι προς την ίδια κατεύθυνση κινούμεθα. Όσον αφορά την απαγόρευση των απορρίψεων, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ο όρος αυτή απαγόρευση δημιουργεί τεράστια υπονοούμενα και δίνει την εντύπωση στον τομέα ότι χρειάζεται να αντιδράσει άμεσα σε εκείνους Φερρυπίν που ζητούν ότι αποτελεί πραγματικά παράλογο αυτό το πράγμα Πρέπει να απαγορεύσουν δηλαδή τις απορρίψεις εκατομμυρίων τόνων ηχθείων στη θάλασσα. Πρέπει να σταματήσουμε, όλοι συμφωνούμε και το έχουμε συζητήσει σε αυτήν εδώ την Επιτροπή επί σειρά ετών, αλλά και ο Αλίας θέλει να του σταματήσει αυτή τη δραστηριότητα. Αλλά ξεχνούμε και αυτοί οι σεφ οι... γνωρίζουν ότι και δεκάδες χιλιάδες μας στέλνουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ότι και οι αλλοίς δεν τους αρέσει να απορρίπτουν αναγκάζονται να το κάνουν αυτό από τι Βρυξέλλε και από το σύστημα διαχείριση το οποίο έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μέχρι τότε να το αναθεωρήσουμε αυτό το σύστημα και μέχρι τότε να βρούμε έναν καλύτερο τρόπο διαχείριση αυτών των αλληλευτικών μα αποθεμάτων, όπω επίση και να κάνουμε αυτό το οποίο έλεγε προηγουμένω ο ομιλητή, να εισάγουμε δηλαδή τεχνικά μέτρα τα οποία θα μα βοηθήσουν στο να αποφεύγουμε να αλλιεύουμε ανεπιθύμητα κάτω του μεγέθου, δηλαδή του επιτροπενού μεγέθου ή εκτό ποσοστώσεων, ήδη Αυτά είναι προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και θέλουμε μέτρα καθημερινής διαχείρισης από τις Βρυξέλλες προς τις περιφέρειες, εκεί δηλαδή τις ελευθερικές ζώνες, προς τα κράτη-μέλη και στην οποία θα συμμετέχουν δηλαδή όλοι οι ενδιαφερόμενοι θέλει, κύκλοι και φορείς, αλλά και οι οι ίδιοι που θέλουν ένα καλύτερο σύστημα, όχι με τόσες πολλές απορρίψεις. Και συμφωνώ επίσης με αυτά που είπατε, ότι θα πρέπει να είμαστε επιλεκτικοί, διότι αν απλώς ζητήσουμε μια πολιτική η οποία θα ισχύει για όλους, θα έχουμε μεγαλύτερη συναισθημότητα, Φερρυπίνη, στον Αστακό, στον Καρχαρία. Αν αρχίσουμε να λέμε στους αλληλείς, δηλαδή, ότι αν κατά λάθο εσείς αλλιεύσετε νέφροπς και αναγκαστείτε να τα εκφορτώσετε, τότε θα αυξήσει την συνεισιμότητα εκθετικά του είδους αυτού. Και αυτό δεν είναι προς συμφέρον κανενός. Επομένως αυτή η ολική απαγόρευση θα πρέπει να εξεταστεί και να σχεδιαστεί και να μελετηθεί. Και πολύ προσεκτικά μάλιστα. Και χαίρομαι για την θέση και τη στάση την οποία λαμβάνετε. Κύριε Λοβέν, παρακαλώ. Κυρία Λοβέν, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την κυρία Ρόντες για την εξαιρετική της παρουσίαση. Και συμμερίζομαι νομίζω πολλές από τις παρατηρήσεις σας και συμφωνώ μαζί τους. Να πω πάντως απευθυνόμενο στην Επιτροπή αυτή γιατί δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, αλλά η Σουηδία, η Δανία και η Νορβηγία προ δύο εβδομάδων δήλωσαν ότι μονομερός, μονομερός θα απαγορεύσουν τις απορρίψεις στο Σκαγεράκι από το αργοτερο απο από 1η Ιανουαρίου του 2013. Το αργότερο. και μιλούμε αυτή μια πλήρη απαγόρευση των απορρίψεων στο Σκαγεράκι. Όχι μόνο αυτών που περιλαμβάνουν στον κατάλογο που βρίσκονται στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ορισμένα είδη δηλαδή και μόνο. Αλλά θα υπάρξει ένας κατάλογος ειδών τα οποία εξαιρούνται όπως καρχαρίες, ή αν θέλετε κάποιες άλλες μέδους του Φερρυπίν που μπορούν να επιβιζήσουν. Αλλά ε, με αυτόν τον τρόπο, αν θέλετε, εφαρμόζεται η απαγόρευση αυτή στην Ορβηγία και λειτουργεί αρκετά καλά το σύστημα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι οι αλληλεί μα είναι σε θέση να γνωρίζουν και γνωρίζουν το πότε δηλαδή και το εάν μπορούν πραγματικά να διατρέψουν τον κίνδυνο να αλλιεύσουν πολλά παραλλιεύματα τα οποία δεν θα έπρεπε. Και αν υπάρξει απαγόρευση των απορρίψεων, ας το, ας το ονομάσουμε έτσι, τότε αυτό νομίζω θα ακυρώσει ούτως ή το πρόβλημα αυτό, θα αποφύγει δηλαδή να αλλιεύουν δηλαδή παραλλιεύματα για τα οποία δεν έχουν ποσόστοση. Θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι οι αλλιείς μας είναι επαγγελματίε. Το σύστημα του πραγματικού κλεισίματος, το επιλεκτικά εργαλεία, Ξέρουμε ότι στη Σουηδία οι αλλιείς χρησιμοποιούν, να θέλετε, αυτά τα εργαλεία επί σειρά ετών, ενώ οι Δανείοι όχι. Και αυτό ήταν η ομολογία του εννοεί, διότι αυτό του συμφέρει. Διότι αν όμω υπάρξει μια απαγόρευση στις αλληλεία, τότε θα έχουμε ίσους όρου ανταγωνισμού για όλου του αλληλεί. Όλοι οι αλληλεί θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα ίδια επιλεκτικά εργαλεία. Και αυτό είναι ο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε την κοινή αλληλευτική πολιτική και στην Ευρώπη, όπου δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν οι ίδιοι όροι ανταγωνισμού για όλου του αλληλεί. Ανησυχώ επίση και για το ζήτημα των απορρίψεων και των ποσοστώσεων απορρίψεων. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο και ένα ερώτημα το οποίο απευθύνεται προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί πολλοί άλλοι λένε ότι αν τώρα οι απορρίψει υπολογίζονται και εκτιμώντα γύρω στο 23% θα πρέπει να αυξήσουμε τι ποσοστώσει μα και τα τάκ μα κατά 23%. Αλλά αυτό θα είναι πολύ και λίγα αντιπαιδαγωγικό ω προ του στόχου τη απαγόρευση των απορρίψεων. Διότι ο στόχο τη απαγόρευση των απορρίψεων είναι να περιορίζεται τα ανεπιθύμητα αλλιεύματα να παραμείνουν αυτά τα ψάρια δηλαδή και τα σποντιλατά στη θάλασσα, εκεί όπου πρέπει να είναι δηλαδή και να μην εκφορτώνονται. Για να μην το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως πρόσχημα για να αυξήσουμε τα τάκια κατά 23%. Και δεν ξέρω ποια είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς αυτό. Τι περιμένετε από το Συμβούλιο επίσης, εσείς Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με ανησυχεί επίσης η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το ταμείο που θα δοθούν χρήματα για να αξιοποιηθούν τα παρελίευματα και να αξιοποιηθούν υποχρησιμοποιούμενα είδη. Αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο τρόπο χειρισμού. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στην επιλεκτική αλία, αποφεύγοντα τα παραλίευματα και όχι να δώσουμε προστιθέμενη αξία στα παραλίευματα, δημιουργώντα έτσι νέε αγορέ για ψάρια τα οποία δεν πρέπει κανονικώ να εκφορτώνονται. Και ένα τελευταίο σχόλιο για τα μεικτά αλλιέματα και το πρόβλημα το οποίο έθεσε η συγκίτρια. Νομίζω ότι θα μπορούσε να ε, λυθεί το πρόβλημα αυτό από τους αλλιείς τους ίδιους, γιατί αν έχουν κάποια ανεπιθύμητα αλλιέματα μπορούν να τηλεφωνήσουν ένα με τον άλλον και αν θέλετε να μοιραστούν αυτά τα αλλιέματα με άλλους. Σύντομη παρακαλώ κύριο Καλτών. Με το σκάνδαλο των απορρίψεων έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κοινή γνώμη. Ξέρουμε ότι είναι ένα νέο πρόβλημα αλλά και μια νέα ευκαιρία που μας προσφέρεται προκειμένου να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο για να αντιμετωπίσουμε ριζικά και όπως πρέπει το πρόβλημα αυτό και το ζήτημα αυτό το οποίο έχει αποκτήσει τεράστιες διαστάσεις από τους κανονισμούς της ε, κοινωτικής αλίας και η άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ξαφνικά δεν είναι απλό το ζήτημα αυτό και ότι μια απαγόρευση των απορρίψεων μέχρι μια ορισμένη ημερομηνία θα λύσει όλα τα προβλήματα. Πολύ απλά το βλέπει και το προσεγγίζει και το αντιλαμβάνεται το ζήτημα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και λάβαμε και ένα σημείο προ λίγων ημερών, το οποίο λέει ότι σε μια μεικτή αλία, που τα πράγματα είναι περισσότερο περίπλοκα, θα πρέπει να υπάρχει το σωστό μείγμα ποσοστώσεων. Αν είναι έτσι απλά τα πράγματα, τότε γιατί, γιατί δεν έχει γίνει και να έχει αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό μέχρι τώρα, ερωτώ. Ε, είναι περίπλοκο, σύνθετο το ζήτημα και βεβαίω αυτό απαιτεί δύσκολες, περίπλοκες και σύνθετες λύσεις. Και χαίρομαι πως η συγγήτρια και άλλοι αναγνώρισαν το γεγονό ότι θα απαιτηθεί και θα πρέπει να δοθούν κίνητρα διότι πιστεύουμε πραγματικά και έχουμε πιστεί ότι τα κίνητρα αν δοθούν θα βοηθήσει και στην επίλυση των προβλημάτων αυτών και κίνητρα που δόθηκαν στην Σκοτία είχαν σαν συνέπεια να μειωθούν σημαντικά και δραστικά οι απορρίψεις βεβαίως με εθελοντική παρακολούθηση, με εθελοντικό κλείσιμο αλληλείας και αυτό οδήγησε σε σημαντική μείωση των απορρίψεων. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Συμβούλιο, στο πρόσφατο Συμβούλιο, απείλησε να αφαιρέσει αυτό το κίνητρο, μειώνοντα τον αριθμό αν θέλετε, των ημερών στη θάλασσα. Αντί του να δώσει και να ανταμείψει μάλλον τους ε, αλείς. Και η Σκοτία βεβαίω είναι ένα παράδειγμα Υπάρχει και το άλλο παράδειγμα ε, που έδωσε προηγουμένω η συνάδελφος, ότι η περιφερειακή, η τοπική απόφαση είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Η Ομοσπονδία των Σκοτε... Σκοτέζων Αλλιέων, όσον αφορά την πρόταση και την απαγόρευση των απορρίψεων, σχολιάζει ότι είναι περίπλοκο το σύστημα αυτό και ότι υπό τις παρούσες προτάσεις υπάρχει ο κίνδυνος οι απορρίψει αυτέ να οδηγήσουν αυτή σε μία ανθρώπινη κατανάλωση. Και αυτό θα είναι εξίσου σκανδαλώδες με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τώρα. Αν επιτρέψουμε δηλαδή να συμβεί αυτό. Αν επιτρέψουμε δηλαδή ένα βρόσιμο ψάρι να έχει αυτή την τύχη. Να μην χρησιμοποιηθεί δηλαδή για ανθρώπινη και κατανάλωση. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο οδηγεί σε απορρίψεις στο πλαίσιο της κοινής αλληλευτικής πολιτικής είναι επίσης όταν υπάρχει και έλλειψη δεδομένων όσον αφορά τα αποθέματα συγκεκριμένων ειδών. Και είχαμε και μειώσει των ποσοστώσεων, πράγμα το οποίο δεν οδήγησε σε μείωση τη θρησιμότητας συγκεκριμένου αυτού είδου, αλλά ε, οδήγησε σε μια αύξηση των απορρίψεων. Περιμένω συνεπώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσει την αναγκαιότητα ότι θα πρέπει από την ε, απλοϊκή αυτή την προσέγγιση ότι τώρα δηλαδή αυτό είναι επιτεύξιμο και εφικτό να γίνει, χωρίς να έχει κάνει κάτι το πολύ σημαντικό και οτιδήποτε να έχει κάνει δηλαδή προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των απορρίψεων. Γι' αυτό λοιπόν να μην βιαστούμε. Ας μην ε, προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε ένα κοινό δηλαδή το οποίο είναι εξοργισμένο πραγματικά αλλά να εργαστούμε και να επεξεργαστούμε ένα σύστημα το οποίο θα επιτυχαίνει δηλαδή το στόχο που είναι η μείωση της νησιμότητος και η μείωση του όγκου των απορρίψεων. Εξασφαλίζοντας ότι θα δοθούν και κίνητρα στα κράτη-μέλη προκειμένου να φροντίσουν να συμβεί αυτό, εγγυόμενο δηλαδή ότι θα αποκομίσουν μακροπρόθεσμα τα ωφέλη από τις θυσίες τις οποίες θα έχουν κάνει μέχρι τότε. Ο επόμενο ομιλητή, πρόεδρε. Αν πρέπει όλες τις απορρίψει αυτές να τις φέρουμε δηλαδή στην ξερά και κατόπιν αποφασίσουμε τι θα τις κάνουμε, τότε κοροδευόμαστε, κοροδευόμαστε, αν πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα έχουμε πετύχει. Διότι θα οδηγήσουμε αυτή σε καταστροφή τον κλάδο τον ίδιο και μετά από πέντε χρόνια δεν θα υπάρχει καθόλου αλία. Έτσι ώστε να εξασφαλίζουν τα προστοζήν όσοι ασχολούνται με την αλία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και νομίζω πως ε, ο όρος δεν είναι σωστός, απαγόρευση των απορρίψεων. Θα πρέπει να βρούμε άλλους όρους, θα πρέπει να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να βρούμε... Θα πρέπει να αποφύγουμε δηλαδή να εκφορτώνονται ε, ψάρια δηλαδή τα οποία είναι πολύ μικρά, δεν τα θέλει δηλαδή η αγορά ούτε και ο καταναλωτή. Και αν το πετύχουμε αυτό τότε νομίζω ότι θα προστατευτούμε και θα είμαστε προστατευμένοι σε σχέση με τις μελλοντικέ εξελίξεις. Δεν πρέπει βεβαίω να υπάρχουν απορρίψει και θέλουμε να καταλήξουμε στην κατάσταση αυτή κάποια στιγμή. Αλλά το πώ θα φτάσουμε εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί όλοι μα Α επισκεφτούμε ένα, πάμε δηλαδή πάνω σε ένα αντιληφτικό για δύο βράδια φερειπίνη, για να δούμε στην πράξη τι ακριβώ γίνεται. Γιατί πολλοί είναι τη άποψη και πιστεύουν ότι όλα αυτά τα αλληλευτικά σκάφη έχουν ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τώρα μπορούμε να πάμε να του πούμε και να πούμε δηλαδή στα, ότι θα πάμε να αλλιεύσουμε δηλαδή εκεί και εδώ και μετά καθώς θα εξαφανιστούμε. Αλλά είναι τόσο γελίο αυτό που δεν πρέπει καν να του δώσουμε την ιαδήποτε αν θέλετε σημασία επί σειρά ετών στον Ηνωμένο Βασίλειο, όταν δεν γινόταν λόγο καν για την ε, απαγόρευση των απορρίψεων, εμεί παίρναμε τα μέτρα μα και τότε ήμουν στο Υπουργείο και ε, ε, συσπίσαμε τεχνικά μέτρα διατήρηση και πρέπει να επισημάνουμε τη σημασία αυτών και να τονίσουμε επίση και τη σημασία του επιλεκτικού εργαλείου και την αποφυγή όλων αυτών. Διότι αν οι απορρίψει, και θα υπάρχουν πάντα απορρίψει, αν εκφορτωθούν, φτάσουν δηλαδή στην ξύρα θα πρέπει να δοθεί ένα κάποιο κίνητρο, θα πρέπει να δοθεί μια κάποια αποζημίωση. Γιατί να πας αν θέλετε στον διευθυντή της τράπεζάς σου και, και να πεις δηλαδή ότι εκφόρτωσα ένα εκατομμύριο απορρίψεις, ο, ο, δεν σημαίνει τίποτα αυτό το πράγμα, ναι, ενώ ο τραπεζίτης θα μπορέσει να στο μετατρέψει και να σου πει ότι τόσο θα αξίζει αυτό σε δίρεση, σε τοπικό νομισμό. μετά από ένα πρόσφατο τηλεοπτικό πρόγραμμα σε ένα από τα κανάλια του BBC. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι πράγμα που ε, προσελκύει, τραβάει. Ε, Αρκούγεται πολύ ελκυστικά. Αλλά πραγματικά καταχρώμαζα και σπαταλάμε δηλαδή πολύ καλά είδου αν θέλετε διατροφής. Και βεβαίως θέλουμε να απαγορευτούν οι απορρίψεις, αλλά τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Και όπως είπε και ο Ιαν, αν ήταν έτσι απλά τα πράγματα, τότε δεν θα υπήρχαν καθόλου απορρίψεις. Ποιος ενδιαφέρεται δηλαδή για να απορρίπτονται αυτά τόσο μεγάλοι όγκοι ψαριών. Όχι οι αλληλείς, θα σου λέω αυτό. Εκείνοι οι οποίοι θα υποστούν τις συνέπειες θα είναι οι αλληλείς οι ίδιοι. Γι' αυτό λοιπόν να αλλάξουμε την ορολογία, τους όρους που χρησιμοποιούμε και ας αλλάξουμε και στάση. Διότι αν δοθούν κίνητρα τότε στην αρχή ενδεχομένω να είναι πολύ δαπανηρά, αλλά σε μεταγενέστερα στάδια θα είναι ιδιαίτερα αποφελή για τις μελλοντικέ γενναίε τα, τα κίνητρα αυτά. Και μην σκεφτόσαστε τι θα γίνει, δεν με ορίζουν, αν θέλετε, τι επόμενε εκλογέ, αλλά σκεφτείτε με ορίζοντα την επόμενη γενιά. Ο κ. Μίλαν. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένα πρόγραμμα ή μια τελόγηση από πλευρά Κομισιών. Υπάρχει ένας ε, κλάδος ο οποίος δεν ε, αρέσκεται πλέον στην ε, στι απορρίψει, αλλά ούτε και η κοινή γνώμη. Αλλά νομίζω ότι η προσέγγιση της Κομισιόν είναι εσφαλμένη. Αντί να ασχοληθεί και να κατανοήσει γιατί το 23% των απορρίψεων θα πρέπει να περιοριστεί, να μειωθεί, ασχολείται με το πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό το 23%. Αυτή είναι μία λάθος προσέγγιση. Από εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε για να μπορούμε να κατανοήσουμε και τις κριτικές που ασκούνται. Θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε το ζήτημα και να δούμε πώς μειώνεται το τμήμα των αλλιευμάτων που αλλιεύεται και είναι αντικείμενο απορρίψεων. Να είμαστε λοιπόν πολύ πιο αυστηροί σε ό,τι αφορά τα εργαλεία αλλίευση και την επιλεκτική αλλίευση αποτελεί μια προτεραιότητα. Είναι θεμελιώδε. Ακόμα, ακόμα και πριν να σκεφτούμε την επίλυση των εκφορτώσεων ή των απορρίψεων. Τώρα, χθε άκουσαμε το μοντέλο Λόβινγκ, το ονομάσουμε έτσι, δηλαδή αυτή την εμπειρία τη Νορβηγία ω μέθοδο. Αλλά και εδώ και θέτω μια σειρά από όλα αυτά θα πρέπει να μην γνωρίζουν όρια σε ό,τι αφορά τι εκφορτώσει. Ή το αλλιεύματα του συγκεκριμένου σκάφου θα πρέπει να σχετίζονται με ε, ε, απορρίψη που επιτρέπονται. Διότι αν δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στα αλλιεύματα και το τι παραλλιεύεται, όντως ε, υπάρχει πρόβλημα χρήσης των εργαλείων αλίας που δεν είναι τα κατάλληλα. Θεωρώ λοιπόν πως εάν δεν εξεδεθεί μια διαφορετική λύση θα πρέπει να υπάρχει σχέση ανάμεσα στα αλλιεύματα και στις ε, εκφορτώσεις ε, της των ενδυνάμει απορρίψεων. Όπως είπα και χθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης ε, της έκθεσης Τρούαν, το ζήτημα του κινήτρου, εάν ο τελικός προορισμός είναι η μεταποιητική βιομηχανία, και ως εκ τούτου υπάρχει μια διτή προσθέμενη αξία, εάν δεν ρυθμίζεται το κομμάτι που συνδέεται με αυτό το σύστημα, τότε πράγματι διακινδυνεύουμε να συμπεριλάβουμε στοιχεία τα οποία θα είναι ίσως και πρόσφορα ή χρήσιμα να αλλιεύονται τα ηχθείς που πρόκειται να απορριφθούν. Λοιπόν, κάνοντας τον ανυπολογισμό των κινήτρων με την τελική χρήση, η οποία θα είναι μεταποίηση, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε ε, μια πολύ πολύ επικίνδυνη business. Και κάτι ακόμα, διότι εμένα μου αρέσουν οι ολοκληρωμένες συζητήσεις, διότι έτσι κομματιαστά η συζήτηση σχετικά με τη μεταρρύθμιση δεν μας βοηθάει και πολύ. Τώρα, δεδομένου του ότι όλα τα λιεύματα εντός ποσοστώσεων που μετά γίνονται εκτός ποσοστώσεων Εγώ φυσικά συμφωνώ με την ε, Ιζαμπέλ ε, η οποία λέει ότι αυτό δεν σημαίνει αύξηση της ποσόστοσης. Δεν θα ίσως να είναι το... να αποτελέσει τον δούριο ύπο και έτσι δεν μπορούμε να δεχθούμε μια πρακτική όταν ε, συζητάμε τις απορρίψεις για να δούμε πώς ε, το Κοινοβούλιο ε, σκέφτεται το ζήτημα των ε, μεταφερόμενων δικαιωμάτων, διότι αυτό είναι ένα κομμάτι ήδη της νομοθεσίας, αλλά δεν θα μπορούσα να πω ότι όντως είναι κάτι το δεδομένο αυτό εγώ, γιατί εγώ είμαι μεταξύ εκείνων που είναι κατά της μεταβίβασης αυτών των αληθικών δικαιωμάτων. Είμαι πεπισμένος λοιπόν ότι αυτά θα πρέπει να παραμείνουν στα χέρια του δημοσίου. Όχι επειδή θέλω το δημόσιο να κατέχει αυτό το αγαθό, αλλά θεωρώ ότι αυτό το δικαίωμα είναι ένα κοινό αγαθό και ως εκ τούτου αυτή της μεταχείρισης θα πρέπει να τύχει. Δεν θα πρέπει να του δώσουμε εμπορική αξία. Λοιπόν, πώς διασυνδέονται όλα αυτά. Υπάρχει κάποια ιδέα, υπάρχει κάποιο σχέδιο στο νου της Κομισιόν. Διαφορετικά όπως έχει το θέμα δεν ε, στέκει. Προτού να ολοκληρώσουμε λοιπόν μια συζήτηση και για τις απορρίψεις θα πρέπει να κατανοήσουμε πώς ε, ολοκληρώνεται το ζήτημα των δικαιωμάτων αλίευσης, διότι τότε ένας πυλώνας ε, του όλου οικοδομήματος γκρεμίζεται και το όλο οικοδόμημα δεν στα στέκει καλά. Η στρατηγική τη Ένωση, λοιπόν σε ό,τι αφορά την μείωση, τον περιορισμό των ε, απορρίψεων λέω ότι είναι ανησυχητική διότι θα χρειαστεί να βρούμε λύσεις ε, ε, την στην μεταρρύθμιση προκειμένου κάτι τέτοιο να μην συμβαίνει. Και φυσικά με, συμφωνώ με τα λόγια του Γκάλαχαν διότι ορισμένα από τα στοιχεία που μας είπε είναι στοιχεία που με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο. Πρόεδρο, θα ήθελα να κάνω και εγώ μερικέ ερωτήσει. Κοιτάξτε, επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε, να πω ότι το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει στις, στις μονοειδής, ε, διότι τα ποσοστώσεις που υπάρχουν υπολογίζονται αναπόθεμα και όχι ανά αλλιεύματα. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα κατανομής και αυτό είναι ένα ζήτημα που υφίσταται διότι δεν έχει αντιμετωπιστεί σωστά. Ο βασικό κανονισμό είχε συμπεριλάβει αυτά τα, δεν είχε συμπεριλάβει αυτές τις ποσοστώσεις και δεν ε, μπορούμε να, δεν μπορεί να υπάρχει προσαρμογή. Τώρα, τα, σε ό,τι αφορά τα παραδιεύματα, θα είναι αυτά τα οποία συμπληρώνουν το πρόβλημα των ποσοστώσεων που έχουν κάποια στις, ε, για τα αλλιεύματα, αυτά τα μονοειδή. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο Και επειδή οι ποσοστώσεις αυτές δεν είναι υποχρεωτικές, είναι, εφαρμόζονται κάτω το πλέον κρατών μελών, δεν μπορούμε να απαιτήσουμε λοιπόν και από τις ε, διοικήσεις ε, να ανταλλάσσουν τα δικαιώματα. Ε, η λύση λοιπόν θα ήταν το ζήτημα, να ρυθμιστεί ζήτημα των παραλιευμάτων. Τώρα, θα έπρεπε κανονικά να είχαμε τελειώσει ήδη, αλλά Βλέπω ότι με κοιτάζετε με φρίκι. Θα σας δώσω 8 λεπτά και θα ζητήσω από τους συντονιστές ε, να ολοκληρώσουμε συντομότερα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα φροντίσω να συμπεριλάβω όλα μέσα σε 8 λεπτά. Καταρχήν, οι ερωτήσεις που τέθησαν να απαντήσω. Οι διατάξει σχετικά με τα είδη που μπορούν να επιζήσουν από την απόρριψη θα μπουν, θα μπουν στον οργανισμό βάσης ή στον οργανισμό ανάπτυξης. Στον οργανισμό ανάπτυξης θα έλεγα, διότι το ζήτημα των απορρίψεων δεν είναι να ε, ε, απαντηθεί ναι ή όχι. Υπάρχουν κάποια είδη που εάν ε, έχουν ε, αλλιευθεί δεν ξέρουμε εάν ε, θα μπορέσουν να επιζήσουν κατά 20, 30, 50%. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί κατά περίπτωση και όπως και οδήποτε άλλο ζήτημα τεχνικού χαρακτήρα θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ρυθμιστεί στον παράγωγο νομοδοσία και όχι στον αρχικό κανονισμό, στο βασικό κανονισμό. Το εάν οι αλληλείς θα πρέπει να έχουν ένα ποσοστό σε παραλογισμάτων σε εθνικό επίπεδο, η Κομισιόν ε, βλέπει με καλό μάτι αυτή την ιδέα. Αλλά έχουμε μια παράδοση ότι δεν θέλουμε να αλλάξουμε, ότι δηλαδή η εσωτερική κατανομή των εθνικών ποσοστώσεων των μελών στου αλληλίστε είναι αποκλειστική αρμοδία του κράτου μέλους. Ωστόσο, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την ιδέα, θεωρούμε ότι είναι θετική, αλλά θα πρέπει να δούμε κατά πόσο το Συμβούλιο δέχεται τα κρατημέλη να έχουν ε, αυτή την υποχρέωση ε, να τις κατανέμουν τις ε, ποσοστώσεις τους σύμφωνα με κάποια στάνταρ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά στα κράτη-μέλη. Εμεί δεν έχουμε πρόβλημα. Τώρα, διάφορε παρεμβάσει ε, αφορούσαν ποσοστά απορρίψεων. Το πρόβλημα που έχουμε είναι περίπλοκο σε, σε μεικτά αλλιεύματα. Δηλαδή, πρέπει να μειώσουμε τα, τις σημαντικά, αλλά ε, το έχει δηλώσει και η Κομισιόν, πρέπει να διατηρήσουμε τη σχετική σταθερότητα. Άρα λοιπόν πώς θα ε, μπορεί να διευθυντηθεί αυτό το ζήτημα. Η ιδέα που προτείναμε είναι ε, πέραν των, ανταλλαγών, των ποσοστώσεων, χρειάζεται να ε, γίνουν αυτές οι ρυθμίσεις όσο γίνεται πιο κοντά στα πραγματικά παραλιεύματα για να γίνει αυτό το είδος των swap. Ε, στην περίπτωση που δεν μπορεί να ρυθμιστεί μερικά το ζήτημα, η Κομισιόν προτείνει αυτές τις ποσοστώσεις, ε, τις συμπληρωματικέ, να τα πάρει το το στόχος στόχο θα είναι στις μεικτά αλιεύματα όπου τα κρατη έχουν μια ποσόστοση μηδενική και δεν πρόκειται καμία μεταφορά δικαιώματο από άλλο κράτο μέλο, αυτό το κράτο μέλο θα πρέπει να έχει το ελάχιστο ποσοστό παραλιευμάτων. Αυτή είναι η, η πρότασή μας και θα πρέπει να συνδυάσουμε τώρα την πολιτική της διατήρησης της σχετική σταθερότητας με αυτήν των παραλιευμάτων τώρα. Όταν ε, θα εξηγήσουμε αναλυτικότερα το νέο δημοσιονομικό αγωνισμό, ε, θεωρώ ότι θα βρεθεί χώρος για να συζητήσουμε το, για το ζήτημα των ταυρίσεων. Τώρα, για περισσότερες ποσοστώσεις για να υπάρξουν διάφο- λιγότερες απορρίψεις, η ιδέα είναι πολύ καλή, είμαστε υπέρ, αλλά μπαίνουμε σε ένα έδαφος που παραδοσιακά ήταν αρμο, της αρμοδιότητας των κρατών μέλων. Θεωρούμε ότι η κοινωνική αρμοδιότητα θα θα υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να εφαρμόζει αυτά τα ποσοστώσει των παραλίευμάτων. Η Κομισιόν δεν έχει πρόβλημα. Θα δούμε κατά πόσο τα κράτη-μέλη είναι διτεθειμένα να παραχωρήσουν κάποια εθνική του αρμοδιότητα. Κύριο Ρομουέβα μίλησε για τον μηχανισμό. Υπάρχουν δύο ζητήματα εδώ. Πώς βλέπουμε την ισορροπία ανάμεσα στην προσπάθεια αποδυνάμωσης των μη επιθυμητών αλευμάτων και δεύτερον τι θα κάνουμε με τα είδη τα οποία δεν επιθυμούμε να αλλιεύσουμε αλλά ε, θα αλλιεύσαμε ούτε ή άλλως, δηλαδή παραλιεύματα. Τώρα η δηλαδη παραλλιευματα συμφωνεί απόλυτα με όλους ε, όσοι δήλωσαν ε, για την ανάγκη βελτίωσης ε, των αλλιευτικών εργαλείων. Φυσικά πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν ποια είναι τα όρια, πού είναι τα όρια. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και αν είχα χρόνο κυρία Πρόεδρε, θα μπορούσα να διευκρινίσω πολλά παραδείγματα σχετικά με τις εμπειρίες που αποκτήσαμε τα τελευταία χρόνια, πώς ένα τεχνικό μέσο που θα βοηθούσε ε, σημαντικά στην μείωση της επιλεκτικότητας και μείωση των απορρίψεων, αύξηση μάλλον της ε, επιλεξιμότητας και μείωση των απορρίψεων ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουν ε, κάποιες δυσκολίες. Ε, πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι ε, δεν μπορούμε να πάμε πολύ μακριά σε ό,τι αφορά την επιλεκτικότητα, δίχως να θίξουμε την οικονομική επιβίωση των στολίσκων. Υπάρχουν περιπτώσεις όπως αυτή των σκαφών της Βορείου Θάλασσας. Μπορούμε να αυξήσουμε την ε, επιλεξιμότητα, να αυξήσουμε τα μάτια στα 120 mm, έτσι θα μειώσουμε φυσικά τα, ε, τις απορρίψεις. Δεν θα μπορούν να ψαρεύουν τότε τα σκάφη αυτά γλώσσα. Αυτός λοιπόν ε, θα ήταν ένα επίτευγμα της αύξησης της επιλεξιμότητας. Ξέρουμε όμως ότι εδώ έχουμε όρια. Δεν μπορούμε να πάμε πολύ μακριά σε κάθε περίπτωση. Εμείς αυτό λέμε είναι να συνδυάσουν πολιτική περιφορά την βελτίωση της ε, επιλεξιμότητας ε, και παράλληλα εξέβρεση μια λύση για αυτά τα είδη που αναπόφευκτο θα συνεχίσουν να αλλιεύονται. Δεν είναι δυνατόν να αποφύγουμε 100% ε, τα παραλιεύματα. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε επίσης είναι να πούμε στον κλάδο. Κοιτάξτε, δεχτείτε αυτή την ε, συμφωνία και αυτά τα ανεπιθύματα αλλιεύματα δεν θα τα, δεν θα πουλάτε, θα τα αφήνετε να σαπίζουν. Λοιπόν, αυτή η πολιτική του να εξευρεθεί μια λύση για το εκφορτωθέν και μη επιθυμητό αλλιεύμα είναι ένα συμπλήρωμα της πολιτικής που θέλει να αποφύγει ε, τα παραλιεύματα, αλλά ξέρουμε ότι ε, μέσω πρόθεσμα δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Θα πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε για αυτά που δεν επιθυμούμε να αλλιεύσουμε, αλλά με όλα τα αυτά, παρά τα αυτά, αλλιεύονται. Και έτσι δεν ναι, θα έλαμε να υπάρχουν εκφορτώσεις ε, αλλιευμάτων τα οποία θα σαπίζουν στα λιμάνια. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε λύσεις, τουλάχιστον μεταβατικές Γι' ε, αυτό είναι το κλειδί της υπόθεση. Θέλουμε ε, μακροπρόθεσμες λύσεις σε ό,τι φορά την επιλεξιμότητα, αλλά τουλάχιστον σε προσωρινό μεταβατικό επίπεδο θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τα είδη τα οποία αναπόφευκτα εκφορτώνονται. Κυρία Λόβιν, όχι δεν θέλουμε να αυξήσουμε τα τάξ, ούτε οι απορρίψει έχουν αυτό το στόχο. Ένα θέμα το οποίο είναι τεχνικού χαρακτήρα θα το προσθέσω το εξηγήσω. Στο τέλος, όπως είδαμε και στο μακροπρόθεσμα προγράμματα, θέλουμε, ο, βασική παράμετρος ε, είναι η θνησιμότητα των ε, ηχθείων. Αν έχουμε λοιπόν ε, ένα κλάδο όπου η θνησιμότητα είναι αυτή που ανταποκρίνεται στην ε, εκφορτωθέντα αλλιεύματα και αυτά τα οποία απορρίφθηκαν. Αυτή η φυσική θνησιμότητα, εάν όλα εκφορτώνονται, θα πρέπει να ισούται με αύξηση του τάκ. Αρκεί να έχουμε σαφής, ε, σαφή υπολογισμό και για τις εκφορτώσεις και για τις απορρίψεις. Δεν θέλουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τις απορρίψεις ως μέσο για να αυξήσουμε τις ποσοστώσεις. Εάν βασιστούμε λοιπόν στη θρησιμότητα αναλύευμα και εκεί όπου γίνεται ένα σωστό υπολογισμό, σωστή μέτρηση, τότε τα τελικά επίπεδα των ποσοστώσεων, των τάξη γνώμη, ε, θα πρέπει να ε, ισούνται με την πραγματική αλλίευση και όχι με αύξηση των ε, τάκ. Δεν θέλουμε να αυξήσουμε λοιπόν τη θνησιμότητα ανά αλλίευμα. Αυτό είναι, αποτελεί κόκκινη γραμμή για μας. Κύριε Χάτστον, να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θέλουμε να ε, παραπλουστεύσουμε τα πράγματα. Θα υπογραμμίσω αυτό που είπε η κυρία Δαμανάκη, ότι για να υπάρξει πρακτική πρόοδο ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα μα υποχρεώνει να καθορίζουμε στόχου ε, μέσω μακροπρόθεσμου για την κατάργηση των απορρίψεων. Πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθούμε όλοι για να βρούμε τις Λύσει ε, που θα μου επιτρέψουν να προχωρήσουμε τώρα. Το ότι η προθεσμία δεν είναι ρεαλιστική, η Κομισιόν έκανε μια πρόταση που θέλει να είναι ρεαλιστική, διότι είναι κλιμακούνται στον χρόνο και το παράδειγμα που αναφέρθηκε εδώ ότι στον Σκαγεράκι δύο κρατημέλη και μια τρίτη χώρα είναι διαιρεθειμένοι να ε, ε, καταργήσουν τι απορρίψει discard ban, Εντάξει, βλέπουμε καλά ότι όταν υπάρχουν τέτοιε πρωτοβουλίε μπορούμε να προχωρήσουμε άμεσα. Ε, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία που αποφάσισαν αυτή την απαγόρευση των απορρίψεων ε, μας κάνουν να πιστεύουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα σε λύσεις. Τώρα για τεχνικά μέτρα, ναι, προτιθέμεθα να ανανεώσουμε τα τεχνικά μέτρα συντήρησης, ε, διατήρησης ε, με μια περιφερειακή προσέγγιση, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν αρχίζουμε να βλέπουμε μέτρα βελτίωση της ε, επιλεξιμότητας αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικής απόδοσης των στολίσκων, και ως εκ τούτου έχουμε κάποιους ε, προφανείς περιορισμούς για το πρόοδο που μπορούμε να πετύχουμε. Δε... απαντώ στην τελευταία ερώτηση, Πρόεδρε, πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το θέμα των παραλυγμάτων. Η ιδέα είναι ότι γνωρίζουμε πως ο στόχος είναι πως σε νυχτές, ε, νυχτά και σε σχετική σταθερότητα τα πολλά κρατημέλη θα έχουν ζήτημα εδώ να επιλύσουν το θέμα. Υπάρχει σχετική σταθερότητα, δηλαδή να προάγουμε και να διευκολύνουμε την ανταλλαγή ποσοστώσεων ανάμεσα τα κράτη-μέλη αυτό είναι ένα μηχανισμό εθελοντικό που μπορεί να επιλύσει τμήμα του, προγράμματος, του προβλήματο, αλλά δεν μπορεί να επιλύσει το σύνολο του προβλήματο σε κάθε περίπτωση. Και αυτέ οι ανταλλαγέ ε, ποσοστώσεων δεν μπορούν να λύσουν το ζήτημα. Γι' αυτό έχουμε προβλέψει ω Κομισιόν ποσοστώσει ε, παραλιευμάτων. Ε, ο στόχο είναι Αν Εάν δύο-τρία κράτη-μέλη έχουν μεγάλη ποσότητα για ένα αλίευμα και καθόλου για κάποιο άλλο, τότε μελετάμε κατά περίπτωση και είναι αυτά τα επίπεδα απορρίψεων αναπόφευκτα, που είναι αναπόφευκτα και προσπαθούμε να βρούμε μια, μια ποσόστοση των παραλίευμάτων σε σχέση με την σχετική σταθερότητα για να μπορέσουν να προσαρμόσουν τα δικαιώματά τους με τις ε, ανάγκες ε, των ε, αδείων. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ όλοι πλην των συντονιστών να εξαφανιστούν ας καρδαμικτή. Por favor, he, he dicho que vayan saliendo todo el mundo que no estén coordinadores. Όσοι δεν είναι συντονιστές, καλούνται να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Παρακαλώ γρήγορα. Σήμερα